Dear colleagues, we are going to start. Αγαπητοί συνάδελφοι. So. Ε, ε, συνάδελφοι, καλημέρα. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Έγκριση τη ημερήσια διάταξης, αν δεν διαφωνείτε. Εγκρίνεται. Um, a few, uh, announcements. Um... Έχω και μερικέ ανακοινώσεις να σας κάνω. Όσοι ήθιστε, διερμηνία διαθέτουμε σε 22 γλώσσες. Έχετε ηλεκτρονικά το φάκελο ε, των εγγράφων. Η δε συνεδρίαση μεταδίδεται ε, ηλεκτρονικά. Δύο πιο ενδιαφέρουσε ανακοινώσει τώρα. Πρώτον, όπως γνωρίζετε ίσως, το μεσημέρι στις 12 έχουμε ε, την πανηγυρική υπογραφή της πολιτικής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2011, ε, παρουσία του Προέδρου ε, Σασόλη και του Γενικού Γραμματέα Κλάους Βέλε. Παρακαλείστε να είστε όσο γίνεται περισσότεροι για να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το γεγονός. Το δεύτερο, αύριο παραθέτουν δεξίωση οι οργανισμοί ε, που συνδέονται με την ΕΝΒΗ στις 12.30 ε, το μεσημέρι. Φυσικά μετά την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεδρίαση. Και θα χαρούμε να δούμε όσο γίνεται περισσότερα από τα μέλη μας αύριο στη δεξίωση αυτή στις 12.30. Ε, προχωρούμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Συστάσεις των συντονιστών έχουν κυκλοφορήσει. Δεν ξέρω, αν δεν έχει διαφωνία κανείς, εγκρίνονται. of the previous... Το, αυτό ισχύει για τα πρακτικά των προηγουμένων συνεδριάσεων. Αν δεν διαφωνεί κανείς, εγκρίνονται. Έχουμε δύο ενημερώσεις σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις, τριμερείς διαλόγους. Το πρώτο ε, αφορά την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Θα σας διαβάσω πού βρισκόμαστε σε αυτό το τριμερή διάλογο. Ε, η δεύτερη συνεδρίαση ε, έγινε. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προχώρησαν στις διαπραγματεύσεις σε, στα δύο πρώτα κλάστερς, ε, την προσέγγιση βάση εκτίμησης κινδύνου και το θέμα των παραμέτρων, παραμετρικών αξιών και ε, παρακολούθησης. Υπάρχουν κάποια θέματα που απομένουν να ολοκληρωθούν σε τεχνικό επίπεδο, ενώ κάποια ευαίσθητα πολιτικά θέματα αναμένεται ακόμα να ε, τύχουν διαπραγμάτευση στις επόμενες συνεδριάσεις. Η πρώτη σύντομη ανταλλαγή απόψεων επίσης ε, έλαβε χώρα συγγνώμη, και ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου δεύτερος τριμερής διάλογος για ένα πλαίσιο ε, που να διευκολύνει την αηφόρο επένδυση. Ξέρετε, αυτό ε, είναι κοινό τριμερής διάλογος Econ. Την πρώτη φορά ε, που συνεδρίασε για αυτό το θέμα, το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο ανέφεραν την εντολή που έχουν το κάθε όργανο, ε, σε σχέση με τα πιο σημαντικά θέματα όπως είναι η σύνδεση αυτού του θέματος ε, με ε, τον κανονισμό για την δημοσίευση των πληροφοριών ε, τους διάφορους δείκτες και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του νέου αυτού κανονισμού ταξινόμησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αντέδρασε στις δηλώσεις ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τόνισε τα σημαντικότερα στοιχεία, ιδιαίτερα τη διακυβέρνηση, διαχείριση και τη θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων. Ο επόμενος τιμερής διάλογος λαμβάνει χώρα απόψε, είναι ο δεύτερος από τέσσερις που προβλέπονται. Προχωρούμε τώρα λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, που έχει ε, να κάνει τη διάσκεψη των συμβαλόμενων μερών COP15. Ε, η συζήτηση θα ακολουθήσει και η προθεσμία κατάθεση απολογιών λίγη αύριο στις 7 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί. Θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στον καθένα ε, στους ε, συνεισηγητές. Η κυρία Ανιές Ευγέν πρώτη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό ε, Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα εκατομμύριο είναι πλέον τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση από τα οχτώ είδη που υπάρχουν στον πλανήτη. Το ένα όγδο των ειδών παγώνει το αίμα μας όταν τα ακούμε αυτό. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι αυτή η άνευ προηγουμένου καταστροφή θα έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στη γη, ε, στην υγεία μας, ε, στη διατροφή, στην υγεία. Η βιοπικιλότητα συμβάλλει στην ποιότητα της ίδιας μας της ζωής και είναι και ένα οχύρο απέναντι στην ε, κλιματική αλλαγή. Ε, η βιοπικιλότητα είναι ε, και εξαιρετική και αναντικατάστατη. Όμως εμείς την ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Ε, είναι ανθρωπογενής η καταστροφή και η διάβρωση που παρατηρείται. Εδώ απέναντι σε αυτή τη διαπίστωση δεν έχουμε πολλά να αντιτάξουμε. Είχαμε βάλει διάφορους στόχους, κανέναν δεν έχουμε πιάσει ούτε τους παγκόσμιους, ούτε τους ευρωπαϊκούς της στρατηγικής για το 2020. Ας μου πει κάποιος αυτό πώς θα το εξηγήσω στους νέους μας. Είναι κατεπήγον η διαφύλαξη της βιοπικιλότητας να γίνει απόλυτη προτεραιότητα, όπως έγινε και η καταπολέμηση της ε, υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό θα πρέπει να φέρει στην Κίνα στο COP15 του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήσει εποχή ε, να είναι συνώνυμο με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε χλιαρούς στόχους που δεν σέβεται κανείς. Θα πρέπει να είναι φιλόδοξοι, μετρήσιμοι ε, και εύκολα αξιολογήσιμη βάση δικτών και μηχανισμών παρακολούθησης. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν και το πνεύμα αυτό αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε αγαπητοί συνάδελφοι και θα συνεχίσω να πηγαίνω σε μια ε, λογική υπερκομματική, διακομματική. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές αλλά και φιλόδοξοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι το πρώτο θεσμικό όργανο της Ένωσης που θα αποφαθεί για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Σέζαρ Λουένα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, το είπε πολύ σωστά η συνεισηγήτρια από το ΕΛΚ. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τον παραλογισμό στην ε, διαφορία και αυτό δεν μπορεί να συμβεί και με το, η σοβαρή κρίση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για τη βιοπικιλότητα. Πάνω από ένα εκατομμύριο ήδη απειλούνται με εξαφάνιση. Είναι αλήθεια, πρέπει να έχουμε φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους, όπως ας πούμε το, τη συμφωνία του Παρισιού θα πρέπει να την, να την κυρώσουμε και να προχωρήσουμε και στην Κίνα στην προστασία της ε, βιοπικιλότητας. Πρέπει να έχουμε περισσότερη φιλοδοξία όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, το 30% του πλανήτη μέχρι το 2030 και το 50% μέχρι το 2050 πρέπει να προστατεύεται. Και εδώ ε, θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες οι σοσιαλιστές. Ε, πρέπει να μιλήσουμε και για την βιώσιμη ενέργεια που μπορεί και πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές ε, μέχρι το 2030 κατά 50% και όλα αυτά ποιος θα τα πληρώσει όχι μόνο οι δημόσιες αρχές, οι πολίτες αλλά και ο ιδιωτικός τομέας και γι' αυτό θα πρέπει να παίξει ρόλο και η φορολογία η πράσινη που θα διέπει ολόκληρο το φορολογικό σύστημα. Θα πρέπει αυτό να εφαρμοστεί όσο γίνεται νωρίτερα, εάν θέλουμε μετάβαση να είναι δίκαιη για όλους και ισότιμη ε, και ώστε να έχουμε μια ποιότητα περιβαλλοντική. Θα πρέπει λοιπόν όσο γίνεται νωρίτερα να μειώσουμε τους, ε, τις εκπομπές για υπέρ της βιοποικιλότητας με δεσμευτικούς στόχους και για την αποψήλωση των δασών, των δασών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει την ευθύνη και έχει, πρέπει να υποβάλει μια, έναν κανονισμό ώστε να δούμε να έχουμε μια αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης με μηδενική ε, ε, επιρροή στα δάση. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τον παραλογισμό στην αδιαφορία σε σχέση με τη βιοπικιλότητα. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you. Uh, for renew, Maria Soraya Rodriguez Ramos. Gracias, Presidente. Bien, como acaba... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως μόλις είπατε, Όπω είπαν όλες οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα και που εργάζονται μαζί μου σε αυτό το ψήφισμα ω συνεισηγητές, βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης εξαιρετικά σοβαρή. Άρα λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε από την τελευταία αξιολόγηση για την βιοπικιλότητα και τις, ε, ε, τα 20, την κατάσταση των οικοσυστημάτων του ΟΗΕ. Αυτό λένε το 66% ε, των διαφόρων οικοτόπων βρίσκονται σε αρνητική κατάσταση και το 88% των ειδών το οποίο παρακολουθείτε μειώνεται ε, διαρκώς στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Γι' αυτό ε, θα πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με μέτρα σοβαρά και διαφορετικά. Άνευ προηγουμένου δηλαδή. Ε, διαφορετικά μέτρα από αυτά που έχουμε κάνει, λάβει μέχρι τώρα σε σχέση με τη βιοπικιλότητα. Να ενισχύσουμε τη διασύνδεση, τη διασύνδεση ανάμεσα στη βιοπικιλότητα και τις ε, περιβαλλοντικές αλλαγές, ώστε να επιτύχουμε ε, ωφέλη και για τις δύο πλευρές, λύσεις που θα βασίζονται στη, βύση, φύση για να διατηρηθεί η βιοπικιλότητα από τη στιγμή που θα έχει μετριαστεί η κλιματική αλλαγή και επίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε χρηματοδότηση κλιματική, κλιματικού τύπου, κατάλληλη όμως για να προστατευτεί η βιοπικιλότητα, ενσωματώνοντας και κινητοποιώντας όλους τους ιδιωτικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για αυτές τις δράσεις. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σε ένα πλαίσιο παγκόσμιο, γενικό, ε, καθολικό και φιλόδοξο και γι' αυτό θα πρέπει εκεί να εντάξουμε με ξεκάθαρο τρόπο μηχανισμούς εφαρμογής, υλοποίησης και αναθεώρησης των λογαριασμών. Προτιθέμεθα να υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες, καθώς και τροπολογίες σε σχέση με τη χρήση των γεών, που επηρεάζει αυτό την, τη χρήση των γιών, επηρεάζει τη βιοπικιλότητα, παίζει σημαντικό ρόλο καθώς και στην ευθύνη που φέρουμε με την κατανάλωση, με τις εισαγωγές και στο πλαίσιο της προστασίας των δασών παγκοσμίω. Πιστεύω λοιπόν πως θα έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο, δεσμευτικό, αλληλέγγυο και καθολικό ψήφισμα. Thank you. Uh, for the Greens. Ευχαριστώ. Βιλενινίστο από τους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο μια επίγουσα κατάσταση στο περιβάλλον, αλλά και για τη βιοποικιλότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, τώρα στο παραπέντε να συμφωνήσουμε επιτέλους για να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτές τις ε, προκλήσεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το κλίμα ε, εξαφάνισης ειδών που είναι ανθρωπογενές, αλλά μπορεί να δημιουργήσει από μόνο του ίσως και μία λύση αν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και παράγουμε τις πρώτε ύλε σήμερα στον κόσμο και στην Ευρώπη. Το χρονοδιάγραμμα είναι πραγματικά πολύ αυστηρό. Η συνάντηση στην Κίνα έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Μα δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και εντό τη Ευρώπη. πρασίνου Μα ικανοποιεί που τα, οι ομάδε στο Κοινοβούλιο θέλουν να αναλάβουν την ηγετική δράση, κυρίω για να, να καλύψουμε και τι επιθυμίε των πολιτών τη Ευρώπη. Έχουμε μια νέα συμφωνία, αλλά δεν είναι αρκετή σε σχέση με αυτό που έχουμε στο σχέδιο. Που θέλουμε μεγαλύτερε φιλοδοξίε, δεσμευτικέ συμφωνίε, καλύτερου στόχου και παγκοσμίω αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλούμε για τι προστατευόμενε περιοχέ. Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα των περιοχών Natura 2000 και να αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματα που έχουν καταστραφεί ή υπονομευθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε καλύτερε ευκαιρίε. Εδώ, έχουμε καλύ... Εδώ έχουμε πρόβλημα γιατί ε, τα μέτρα που έχουμε δεν προχωρούν σωστά. Πρέπει να ε, έχουμε μεταρρυθμίσει. Η βιοπικιλότητα, ωστόσο, δεν βρίσκεται πολύ ψηλά στι μεταρρυθμίσει που πρέπει να κάνουμε στην, στην κοινή γεωργική πολιτική. Η δασοκομεία, ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε πιο ψηλά και την βιοπικιλότητα, γιατί η κατάσταση πραγματικά δεν μειωμένη. Πρέπει λοιπόν έτσι να ε, συμβάλλουμε και στην προστασία των ε, ειδών, τα οποία σύμφωνα ε, με τα επιστημονικά δεδομένα μπορεί να οδηγούν και στην απώλεια βιοπικιλότητας. Εδώ έχουμε το θέμα επίσης της χρήσης των γεών και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε στην Κίνα όταν θα πάμε στην ΚΟΠ. Η αποψήλωση των δασών επίσης, η απερίμωση είναι Σημαντικό θέμα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε προοδευτικοί εδώ για να μπορέσουμε να έχουμε ένα παγκόσμιο στόχο και για αυτό στην Κίνα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε στην ECR. Ε, Αλεξάνδρ Βόντρα. Πες το αυτό για τη Χάιντι. δεν έχει υπογράψει το ψήφισμα όμως. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ECR είναι ε, δεσμευμένη και αφοσιωμένη στο να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Η προστασία της βιοποικιλότητας, θεωρούμε ότι είναι πολιτική μας ευθύνη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι πρέπει να δράσουμε. Οι επιστήμονες ε, μας ε, προειδοποιούν ότι ένα εκατομμύριο ήδη απειλούνται με εξαφάνιση και η επόμενη ε, συνάντηση CBD του χρόνου θα είναι πραγματικά σημαντική για τα αποτελέσματα για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Υπάρχουν λόγοι λοιπόν που πρέπει να δράσουμε. Κάποιοι από τους στόχους για την βιοποικιλότητα δεν ε, θα επιτευχθούν μάλλον μέχρι το 2020. Και διακινδυνεύουμε να αποτύχουμε, διακινδυνεύουμε να υπάρξει μεγάλη υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Πρέπει να απαντήσουμε βεβαίω και σε κάποια ερωτήματα και για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και για τα πολιτικά κόμματα στην COP15, ε, όπως ας πούμε το πώς θα διατηρήσουμε τις φιλοδοξίες με τους νέους στόχους, ενώ θέλουμε ταυτόχρονα να προωθήσουμε επιτόπου δράσεις, ε, πώς θα μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε και με άλλους παγκόσμιους στόχους και με τους στόχους του ΟΗΕ, οι νέοι στόχοι πώς θα συνδεθούν με τις, ε, δεσμε... με τις δεσμεύσεις για την μεταφορά τεχνολογίας, για τη δημιουργία ικανοτήτων, για τα οικονομικά θέματα, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και τέλος πώς ε, μέσα στα πλαίσια του πλαισίου CBD μπορούμε να ε, διατηρήσουμε τις νέες τεχνολογίες και τα στοιχεία τα επιστημονικά. Σίγουρα το ψήφισμα αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό σημείο κίνησης. Θα υποβάλουμε τροπολογίες έτσι ώστε να έχουμε τελικώ ένα πολύ καλό κείμενο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την επικοδομητική συνεργασία με άλλους ε, σπόνσορες έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σίλβια Μόντικ για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους προηγούμενους ομιλητές. Χαίρομαι που υπάρχει η υπερκομματική στήριξη, γιατί δεν μπορούμε να το τονίσουμε επαρκώς το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, τα στοιχεία που έχουμε για τη βιοπικιλότητα, για τα διάφορα είδη που απειλούνται, που βρίσκονται στο σημείο της εξαφάνισης, είναι πραγματικά τρομακτικά. Η βιοπικιλότητα πραγματικά υποφέρει όπως υποφέρει και το κλίμα. Και Έχουμε έναν στόχο που θέλουμε να τον πετύχουμε μέχρι το 2020, αλλά πρέπει να πάμε και επέκεινα. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί νέα μέτρα, μια νέα στρατηγική. Αλλά τι νέο έχει τελικώ αυτή η στρατηγική. Είναι σαφέ ότι αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετά. Χρειάζεται νέα μέθοδο, χρειάζονται νέε ιδέε, χρειάζονται μετρήσιμοι στόχοι, χρειάζονται πιο δεσμευτικοί στόχοι. Και χρειάζεται επίσης και νομική παρέμβαση, νομική ισχύς. Η γεωργία και η δασοκομεία είναι ούτως ή άλλως ένα κομμάτι της εξίσωσης. Η υποβάθμιση της βιοπικιλότητας ε, είναι σημαντική και πολλές φορές και κυρίως στη χώρα μου ε, οφείλεται στην ε, δασοπονία. Ε, θα μπορούσαν οι κανόνες να είναι πιο αυστηροί. Η γεωργία πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βοηθήσει, να προστατευτεί η βιοπικιλότητα. Πρέπει να επιτύχουμε τους ε, στόχου που έχουμε θέσει, πρέπει να επιτύχουμε του στόχου τη Συμφωνία του Παρισιού, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση τη βιοποικιλότητας. Ελπίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή ΕΝΒΗ θα εμπλακεί και στο μέλλον της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής, γιατί ε, δυστυχώς εάν ακούσουμε μόνο τους, ε, το λόμπι της δασοκομείας και της γεωργίας, δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε μια καλή και φιλική προς το περιβάλλον γεωργική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Catch the eye τώρα. Πριν να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. That's it. Okay, so I think there are more. So we start with Klaus Birner for the Greens. Εμένα εννοείται πρόεδρε. Ωραία. Για την αντιμετώπιση της, των προβλημάτων στη βιοπικιλότητα. Θεωρούμε ότι οι κότοποι για τα ζώα και τα φυτά μειώνονται. Και βεβαίως συνήθως τα εντομοκτώνα και τα διάφορα δηλητήρια είναι υπεύθυνα. Αυτό που ξεχνούμε ωστόσο είναι ο αντίκτυπος ε, των, της ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας ε, και ακτινοβολίας. Έχουμε δει έρευνες για τους μηχανισμούς και τον αντίκτυπο και ξέρουμε πώς βλάφτει αυτή η ακτινοβολία. Αλλά δεν το λαμβάνουμε υπόψη γιατί έχει, κρύβονται πολλά οικονομικά συμφέροντα πίσω από αυτή. Μπορούμε να το δούμε αυτό και στα δέντρα και κυρίως τα τμήματα των δέντρων που ε, ε, ακτινοβολούνται καταστρέφονται, πεθαίνουν μετά από 2-3 χρόνια και όσα δεν βρίσκονται σε ζώνη ακτινοβολίας και παρόλο που όλα βρίσκονται στο ίδιο δέντρο και ε, ποτίζονται με το ίδιο νερό δεν παθαίνουν τίποτα. Το ίδιο παρατηρούμε και στα ζώα. Οπότε παρακαλώ επιγόντως και αυτόν τον βλαβερό μηχανισμό που, οφείλει, που βοηθά στην ε, καταστροφή των ειδών να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ για αυτό το ψήφισμα πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε αισθητή, ε, σαφή τη φωνή του Ευρωκοινοβουλίου. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε κάποιες πτυχές που πρέπει να ενισχυθούν στο εσωτερικό του ψηφίσματος για ε, να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε και να τονίσουμε πόσο επίγουσα ε, είναι μια ρηξικέλευθη αλλαγή και μια ουσιαστική πολιτική γιατί εδώ και καιρό ξέρουμε πως η συσχέση συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην ευθροπινή δραστηριότητα και την άνευ προηγουμένου μείωση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε πια να αρνούμεθα, να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να το αγνοήσουμε και να μην το αντιμετωπίσουμε, γιατί ε, όχι μόνο σε Ευρώπη, σε παγκόσμιο επίπεδο θα επιτύχουμε τα, τους στόχους του 2020, αλλά οι νέες σχέσεις μας επιβεβαίωσαν το Μάιο ότι με το ρυθμό αυτό της απώλειας της βιοπικιλότητας έχουμε τεράστια και δραματικές, δραματική επιρροή σε, ακόμα και στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ας πούμε, ε, ε πείνα, φτώχεια, ωκεανοί, γέες, ε, ακόμα αυτοί που είναι φτωχότεροι είναι αυτοί που θα πληγούν και περισσότερο. Είναι λοιπόν άνευ προηγουμένου και διαρκώς αυξάνεται ο κίνδυνος απίστευτος ο αριθμός του ενός εκατομμυρίου ειδών που μπορεί να εξαφανιστούν για πάντα. Είναι σωστό σημαντικό ε, αυτό το Ευρωκοινοβούλιο να δεσμευτεί με ένα ψήφισμα όσο γίνεται πιο φιλόδοξο, ώστε η Ευρώπη να εγκαταλείψει οριστικά τη λογική της εθελοντικής δέσμευσης και να προχωρήσει προς δεσμεύσεις που να είναι υποχρεωτικές, δεσμευτικές και ε, σημαντικές για την επίτευξη των στόχων. Πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης ξεκάθαρος μέχρι το 2030 με σαφείς δείκτες απόδοσης και διαφανεί ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε τις ευθύνες σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο ως πολίτες. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ από την ομάδα Renew ε, Europe. Η κυρία Σαμπό. Πρόεδρε, συμφωνούμε νομίζω όλοι στις διαπιστώσεις για τη βιοπικιλότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή ολόκληρη στον πλανήτη, για τους ε, πληθυσμούς γενικότερα. Θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτές τις λύσεις που βασίζονται στη φύση, στα χερσαία, ε, θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα να θεωρηθεί τμήμα της λύσης και όχι του προβλήματος και της λύσης καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Υπόθηκε επανειλημμένα. Θα πρέπει να μας προβληματίσει περισσότερο αυτή η ιδέα που προωθεί η Διεθνής Ένωση για τη Διαφύλαξη της Φύσης να τιμολογηθεί κάπως η φύση. Τι εννοώ. Κάποιος αναφέρθηκε στη συνοχή που θα πρέπει να χαρακτηρίζει για τη συνέπεια τις πολιτικές μας. Εμείς μιλήσαμε προηγουμένως για τις αλλάσεις μεταφορές, αλλά μόνο για τις εκπομπές. Τι γίνεται όμως για τον αντίκτυπο ε, ε, των κινητήρων των πλοίων ε, στη βιοπικιλότητα. Κινητήρες που είναι σε λειτουργία όχι μόνο εμπλό, αλλά και στους λιμένες. Επίσης, η βιοπικιλότητα είναι κοινό αγαθό για όλους δεν είναι μόνο υπόθεση των κρατών, των συλλόγων, των γεωργών, των ναυτικών, των ε, βιομηχανιών, αλλά όλων των πολιτών. Και θα πρέπει να γνωρίζουν όλη τη βιοπικιλότητα. Είναι ευθύνη όλων μας. Θα πρέπει να προωθήσουμε επίσης ε, αυτή την ιδέα της συμμετοχικής επιστήμης. Ε, δηλαδή να υπάρχουν κάποιες δράσεις και από για ενημέρωση για εκπαίδευση, όπως είναι κάποια θαλάσσια πάρκα που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ από τους Πρασίνους. Η κυρία Πάουλους. Ευχαριστώ. Στα αγγλικά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα. Κοιτάξατε τη μελέτη που έκανε το Ινστιτούτο της Στοχόλμης για την ανθεκτικότητα θα διαπιστώσετε ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή ο φόσφορος και ε, το άζωτο απειλούν τα εδάφη και ε, τα ύδατα. Και γι' αυτό από μόνο απειλείται η βιοπικιλότητα. Γιατί Υπάρχουν φυτά και ζώα, δηλαδή χλωρίδα και πανίδα, που είναι συνηθισμένα να ζουν σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις υδρογόνου, ε, συγγνώμη, αζότου και φωσφόρου. Ε, αυτό λένε οι οικολόγοι, ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Πριν φτάσουμε ακόμα στα φυτοφάρμακα. <coughs> Uh, αν δεν απατώμε, ε, δεν υπάρχει ε, άλλος συνάδελφος που να έχει ζητήσει το λόγο στο Catch οπότε μπορούμε να περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας που συζητά αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Όντω ε, είναι θέμα οικολογικής κρίσης αυτό που συζητούμε, που ξεπερνά την ε, ε, κλιματική αλλαγή και βεβαίω απειλεί την ύπαρξή μας, την βιόσφαιρα που εξαρτάται από, το τι από την οποία εξαρτώμεθα. Και βεβαίω έχουμε δει ότι όντω αυτό είναι ένα από τα όρια που σχετίζονται και με τον ε, κύκλο των θρεπτικών συστατικών. Αυτό που γνωρίζουμε για την COP15 ε, που ε, έρχεται είναι ότι θα, μπορεί αυτό το, θα πρέπει αυτό το νέο σύστημα να είναι καινούριο, θα πρέπει να είναι θεμελιώδες και γι' αυτό, αυτό μάλιστα μας λένε και οι επιστήμονες. Έχουμε το διακυβερνητικό πάνελ ε, για, τα, ε, για τις υπηρεσίες που είναι ξεκάθαρο και λέει ότι όντως είμαστε, ε, υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε ένα εκατομμύριο είδη εάν συνεχίσουμε τα πράγματα όπως έχουν. Και βεβαίως έχουμε καταγράψει και τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην απώλεια βιοποικιλότητας. Ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι οι παράγοντες. Η χρήση, η υποβάθμιση της γης καταρχάς η υπερβολική εκμετάλλευση των γεών και των ωκεανών, η κλιματική αλλαγή από μόνη τη, η μόλυνση διαφορών ειδών και τα ανθεκτικά είδη. Δεν είναι λοιπόν κάτι συνηθισμένο αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτού του συγκεκριμένου παράγοντε. Στι πολιτικέ κατευθυντήρες γραμμέ τη ε, νέα Προεδρού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν πολλά που αναφέρονται στο κλίμα και στην ανάγκη που υπάρχει να είμαστε οι πρώτοι ουδέτεροι προ τον άνθρακα ήπειρο ε, στον κόσμο. Και Βεβαίω, κατά την άποψή μου, τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι καινοφανή. Πρέπει να ε, αποκαταστήσουμε τα συστήματά μα. Αυτό πρέπει να καθοδηγεί τη δουλειά που θα γίνει. Η βιοπικιλότητα, η υποβάθμιση τη γη, τα τρόφιμα, όλα πάνε χέρι-χέρι. Χρειαζόμαστε νέα πρότυπα για την βιοπικιλότητα στι βασικέ πολιτικέ από τη γεωργία, τη βιομηχανία, την δασοπονία, την οικονομία και κυρίω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει την ηγετική δύναμη σε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο όπως υπάρχει για το κλίμα. Γι' αυτό όταν μιλούμε για το ποια θα πρέπει να είναι τελικώ για το 2030 η νέα ε, στρατηγική, η οποία αναφέρεται και στην Πράσινη Συμφωνία, στο Green Deal, θα πρέπει να έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ένας που θα ασχολείται με, το, με την ε, Ευρωπαϊκή Παρέμβαση για το Παγκόσμιο Πλαίσιο που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2050 αλλά και για τους στόχους που έχουμε θέσει και τα ορόσημα για το 2030 αλλά κυρίως για το πώς μπορούμε να ε, δείξουμε το ότι είμαστε υπόδειγμα, πώς μπορούμε να, ε, έχουμε κάποιες δεσμεύσεις για να αντιμετωπίσουμε τις, την απώλεια της βιοπικιλότητας. Πολλοί το είπαν στις παρεμβάσεις τους Μία από τις πτυχές που λείπει σε ό,τι αφορά την πολιτική για τη βιοπικιλότητα είναι η έλλειψη της ε, μετρησιμότητας, της ποσοτικοποίησης. Είναι εύκολο να μετρήσει κανείς το ε, διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από την ε, απώλεια της βιοπικιλότητας, αλλά η επιστήμη προχωρά. Και υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες τώρα να έχουμε ποσοτικούς, ποσοτικοποιημένους στόχους και βεβαίως πρέπει να έχουμε και ένα συνολικό στόχο ως προς αυτό, έτσι ώστε να μας βοηθήσει να φτάσουμε και στο, όπως μας βοηθά για την μείωση κατά 1,5 βαθμό για την θερμοκρασία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το προωθήσουμε. Δεύτερον, για την βιοποικιλότητα και την πολιτική είναι το ότι δεν υπάρχει βασικό mainstreaming, δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση και ε, εφαρμογή των δεσμεύσεων σε βασικές πολιτικές. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Να αναφερθώ σε κάτι που αναφέρθηκε σε αρκετές παρεμβάσεις των μελών η βασική σύνδεση με, τις, με την κλιματική αλληλεγγύη. Δεν μιλούμε για δύο ξεχωριστά θέματα εδώ, προβλήματα. Μπορούν το ένα να βοηθήσει ή να ε, υποβαθμίσει το άλλο. Και υπάρχει μάλιστα και μεγάλη δυνατότητα να έχουμε ένα πολύ καλό και θετικό πολιτικό μήνυμα για τις ε, λύσεις που μπορούμε να προβλέψουμε. Δεν είναι δηλαδή ένα έξτρα βάρος. Η αποκατάσταση της φύσης μπορεί να δώσει πολλά ωφέλη για τους ε, και να βοηθήσει φυσικά και στην κλιματική αλλαγή. Οπότε θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα ε, οριζόντια σε όλε τι πολιτικέ και να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι βασικέ πιέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είμαστε εμεί το παράδειγμα για το τι πρέπει να γίνει σε διεθνέ επίπεδο και σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των κονδυλίων, την συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων αλλά και να εξασφαλίσουμε για τη βιοπικιλότητα δίκαιη μετάβαση για όλους όχι μόνο για τα ορυκτά καύσιμα, ας πούμε, αλλά γενικώ για τον τομέα τη βιοπικιλότητα που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις, ε, σε όλε τι πολιτικέ με δίκαιο τρόπο. Το ξαναείπα. Ε, χρειαζόμαστε ένα θετικό μήνυμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή ε, μόνο αντιμετωπίζοντας την εξαφάνιση που έχουμε προκαλέσει. Πρέπει να βασιστούμε και σε κάποιες αξίες για τη φύση και για την ομορφιά της φύσης. Πρέπει να, πρέπει να τη διατηρήσουμε. Αλλά αυτή η αξία και τα ωφέλη που μπορεί να έχει κανείς με, με, τη, μέσω της διατήρησης της φύσης για την οικονομία, για, την, για το περιβάλλον κτλ. Η δουλειά που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πραγματικά πολύ καλή. Τονίζει τον επίγοντα χαρακτήρα, τονίζει τη διασύνδεση με, τις, με τη γεωργία, με την κλιματική αλλαγή, με τη χρηματοδότηση. Αν μπορώ να προτείνω κάποιους τομείς που θα μπορούσατε ίσως να μελετήσετε, θα αναφερθώ σε κάποια από τα σχόλια των μελών σας. Ας πούμε το θέμα της, ε, του αποτυπώματος της βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σύνδεση με την κατανάλωση και το εμπόριο. Επίσης, οι ε, στόχοι για τις προστατευόμενες περιοχές και τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ίσως εκεί να είναι πιο εύκολο να έχουμε ποσοτικοποιημένα στοιχεία. Επίσης, έχουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για την ενίσχυση των δράσεων για την προστασία των δασών κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια, μια σύνδεση και με την Συμφωνία του Παρισιού. Αλλά βεβαίως εδώ θα πρέπει να δούμε και την ε, σύμβαση της ε, βιοπικιλότητας, η οποία επίσης έχει κάποια εργαλεία, ίσως να μην είναι επαρκή, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ ένα νέο σκεπτικό εθνικής παρέμβασης, αφοσίωσης για την αντιμετώπιση του κλίματος για να ενισχυθούν δηλαδή και οι εθνικές στρατηγικές για τη βιοπικιλότητα και τα εθνικά ε, σχέδια τα οποία μπορούμε να τα συνδέσουμε με ε, ε, επαληθεύσιμους στόχους και ποσοτικοποιημένα συστήματα. Επίσης, η χρηματοδότηση. Να σας προειδοποιήσω εδώ για κάτι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέε δομέ με νέα κονδύλια, όταν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπάρχοντα, όπω το Παγκόσμιο Ταμείο πούμε, για, την, για το περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσαμε να εντάξουμε τα θέματα της βιοποικιλότητας. Δεν θα πω άλλα για το τι άλλο χρειάζεται να καλυφθεί. Σας παραπέμπω και στο ε, κείμενο που έχετε καταγράψει και ελπίζω ότι το ψήφισμα αυτό όντω θα είναι πολύ καλό κείμενο για να μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Θα δούμε βεβαίω τι θα περιλαμβάνει, τι μηνύματα θα έχει το ψήφισμα αυτό. Για τη διαδικασία τώρα. Λοιπόν, τι κάνουμε από εδώ και μπρο. Έχουμε την ε, προθεσμία για τι ε, τροπολογίε, όπω είπα, αύριο στι 11. Ψηφοφορία στην ΕΜΒΙ Δεκέμβριο στι 2 ή στι 3, στην επόμενη σύνοδο. Και μετά, θα το επιβεβαιώσουμε βεβαίω, έχουμε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Και παραλλήλως βεβαίως ε, έχουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία περιμένουμε, τα οποία μπορεί να έχουν ίσως εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους ή μέχρι τις αρχές του επόμενου. Άρα το ψήφισμα αυτό θα είναι η πρώτη ευκαιρία ή ίσως και η τελευταία ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμως να λάβει θέση πια ε, για, την, ε, για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και για την εντολή που απορρέει από την Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα. Είναι βεβαίω πολύ σημαντικό το ψήφισμα αυτό για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Οπότε νομίζω ότι αυτή η συζήτηση κλείνει και μπορούμε να πάμε στο επόμενο θέμα σε ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ θα γίνει τώρα μια κοινή συζήτηση για τα θέματα από το 7 έως και το 10 για τις αντιρρήσεις σχετικά με διάφορα θέματα γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ε, θα δώσω το λόγο στους βουλευτές που υπέγραψαν ε, το σχέδιο ψηφίσματος ε, τη Μέτς από τους Πρασίνους και μετά ε, σοσιαλιστές, πράσινους, μία γεγραμμένους στη ΣΥΡΠΑ, είναι και στους υπολείπους ε, που θέλουν να μιλήσουν βουλευτές και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μέτς από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εδώ είμαι. Ε, τέσσερις αντιρρήσεις έχουμε για τέσσερα γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που έχουν καταστεί ε, σε ένα ή περισσότερα φυτοφάρμακα και μεταξύ αυτών και η γλυφοσινάτη και η γλυφοσάτη. Ε, επ' ευκαιρία της συζήτησης λοιπόν θέλω να ρωτήσω τρία πράγματα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαπίστωσα ότι συχνά διαφωνούμε ε, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, για, μάλιστα ε, για το τι ισχύει Συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αποφασίζει θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε νομοθεσία και διάφορους θεμητούς ε, παράγοντες. Ε, δεύτερον, Ποια είναι, ποιοι είναι οι θεμητοί παράγοντες. Η προστασία της βιοπικιλότητας είναι αθέμητος παράγον. Η αυξημένη έκθεση σε τοξικά φυτοφάρμακα δεν είναι θεμητός παράγον για αγρότες σε τρίτες χώρες η μεγάλη αποψήλωση των δασών ευρείας κλίμακας δεν είναι θεμητός παράγων. Τώρα περιμένω ότι θα μας πείτε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ε, στην διακριτική ευχέρεια και ευθύνη των τρίτων χωρών. Εμείς όμως ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υπογράψει διεθνείς συμφωνίες και για το περιβάλλον. Συμφωνεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλή ερώτηση ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το περιβάλλον όπως είναι η Συμφωνία των Παρισιών και άλλες, όταν εγκρίνει αδειοδότηση κυκλοφορίας ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ευχαριστώ. Γκίντερ Σίδλ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Αξιότιμοι συνάδελφοι, σε αυτό ε, το ψήφισμα που ψηφίσαμε εδώ στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια, ε, είχαμε πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο και σήμερα. Ε, το απόγευμα να επαναληφθεί. Πρόκειται και για νέες άδειε, αλλά και για παράταση ε, άδεια για γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι, δύο είδη αραβοσίτου και ένα είδος σόγιας. Ε, έχουμε, ε, έχουμε δει ότι έχουν γίνει ανθεκτικά αυτά, μία φορά οι περισσότερες για φυτοφάρμακα και ειδικά στον αραβόσιτο υπάρχει ένα γονίδιο το οποίο είναι τοξικό για διάφορα έντομα και για προνύμφες. Ε, γλυφοζινάτη και γλυφοζάτη. Ε, το γλυφοσυνάτη ε, θεωρείται ότι βλάπτει το αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου και από την 1η Οκτώου το 2018 απαγορεύεται και ενδεχομένω είναι και καρκινογόνες κάποιες ουσίες αυτές και γίνεται και έρευνα. Απαγορεύονται στην Αυστρία Και αυτό είναι ενδεικτικό και υποστηρικτικό αυτή της άποψη. Ε, μια που τα είπα όλα αυτά, θέλω να τονίσω και πάλι ότι η καλλιέργεια μεταλλαγμένων φυτών οδηγεί σε μεγαλύτερη χρήση φυτοφαρμάκων και δημιουργούνται αντοχές και ε, σε άλλα είδη και αυτό οδηγεί σε περισσότερα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στις οδιές. Αν στην Ευρώπη συζητούμε μέτρα ή αποφασίζουμε απαγόρευση ε, δηλητηρίων και φυτοφαρμάκων από τη μια και από την άλλη εισάγουμε προϊόντα ε, που ανθίστανται στα φυτοφάρμακα, αυτό δεν είναι αντιφατικό. Κατά την άποψή μου είναι και συνεπές. Γι' αυτό οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, η δική μου πολιτική ομάδα, θα καταψηφίσει ε, αυτή την πρόταση. Δηλαδή θα υπερψηφίσει την αντίρρηση η Άνια Χάζεκαμπ από την ΚΟΕ. Ε, δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίνει νέες ε, άδειες και παρατείνει τις παλιές για τη σόγια, τον αραβόσιτο και το βαμβάκι. Αυτά και βλαβερά είναι και δημοκρατική νομιμότητα δεν έχουν και θα αυξήσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων επικίνδυνων. Αυτή η αρχαϊκή καταστροφική ε, γεωργία είναι κάτι το οποίο πρέπει να εγκαταλείψουμε αν θέλουμε να έχουμε μία πιθανότητα να σώσουμε το πλανήτη. Και μάλιστα αυτά τα είδη που είναι ανθεκτικά σε γλυφοσινάτη και γλυφοσάτη που είναι δηλητήρια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ε, παράγουν και τοξίνες ε, BT που βλάπτουν τις πεταλούδες και διάφορα έντομα. Αυτά είναι του προηγούμενου αιώνα, όταν θεωρούσαμε ότι τα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα είναι η λύση και τώρα ξέρουμε όμως ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα. Επίσης γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βγει να μας πει ότι είναι υποχρεωμένη να εγκρίνουν αυτές τις εισαγωγές ακόμα και αν δεν υπάρχει ποτέ ε, ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών υπέρ της έγκρισης. Δεν ισχύει αυτό. Βεβαίως ε, δεσμεύεται νομικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Προσφυγών, αλλά το άρθρο 6 παράγραφος 3 ε, του κανονισμού της Επιτροπολογίας επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προβεί σε αυτή την έγκριση αν δεν υπάρχει πλειοψηφία των κρατών μελών που να συμφωνούν. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί την εκτίμηση της ΕΦΣΑ, ιδιαίτερα όταν δεν είναι πλήρης και δεν συμπεριλαμβάνει ε, τα κατάλοιπα αυτά τα επικίνδυνα των φυτοφαρμάκων. Ε, απλή ερώτηση λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους θα δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να ε, διοδοτήσει άλλα μεταλλαγμένα αν δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε για να σεβαστείτε τη δημοκρατική λήψη των αποφάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Λεωνόρα Εύη, από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μεγάλη πλειοψηφία των γενικώ τροποποιημένων οργανισμών και που, είναι, που εισάγονται έχουν ε, αντίσταση σε πολλά φυτοφάρμακα. Βεβαίως ε, υπάρχει μείωση των καταλήπων στις εισαγωγές, αλλά τα, τα υποπροϊόντα όλων αυτών ε, έχουν πραγματικά σουρευτικό αντίκτυπο και ε, εκπίπτουν του πάνελ ε, των γενετικών σωροποιημένων της ΕΦΣΑ. Όπως έχει αναγνωρίσει λοιπόν και η ΕΦΣΑ, ο τρόπος με τον οποίο τα ζανιοκτώνα επιβαρύνουν τις ε, καλλιέργειες ε, μπορούν να οδηγήσουν σε ε, επιπλοκές για την τοξικότητα των ουσιών. Οπότε, πότε και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή <laughs> προτίθεται να κλείσει αυτό το κενό στην αξιολόγηση κινδύνου, έτσι ώστε τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων να αξιολογούνται επαρκώς στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Πιετικάινεν. Ε, έχει ζητήσει να μιλήσει αλλά δεν είναι εδώ. Οπότε δίνω το λόγο στο ΕΛΚ. Thank um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επαναλάβω κάποια από, αυτά που έχω ξαναπεί στην Επιτροπή που την τελευταία φορά που συζητούσαμε αυτά τα θέματα και παρόμοιες αντιρρήσεις γιατί η γραμμή του ΕΛΚ δεν έχει αλλάξει από τότε. Νομίζω ότι η ΕΦΣΑ έχει δώσει αυτή την εντολή, δεν την έχουν ξεπεράσει και το ερώτημα που τίθεται είναι ότι τελικώς δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε την γνωμοδότησή της. Αλλά αφού δεν την ε, ε, χρειαζόμαστε, αφού δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την γνωμοδότησή της, τι χρειαζόμαστε την ΕΦΣΑ όλος διόλου σε πολλές περιπτώσεις ε, δεν έχουν ε, καταγράψει κάτι που να δείχνει ότι αυτά, αυτές οι καλλιέργειες είναι πολύ πιο βλαβερές από τις πιο συμβατικές και νομίζω ότι η ΕΦΣΑ λέει ότι το προϊόν είναι ασφαλές. Άρα αφού λέει ότι είναι ασφαλές πρέπει να ε, συμφωνήσουμε να δεχτούμε την επιστημονική της γνώμη. Θεωρώ λοιπόν ότι η Κομισιόν δεν έχει υπερβεί την εντολή που έχει και εγώ θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους να ε, καταψηφίσουν αυτήν την αντίρρηση. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανένα το λόγο από την Renew, οπότε πάμε στην ECR. Αλεξάνδρ Βόντερ. Ευχαριστώ. Πριν ε, δύο λεπτά συζητούσαμε την ε, βιοπικιλότητα και ήμασταν τυχεροί γιατί η ιδεολογία και η επιστήμη βρίσκονται στο ίδιο, στην ίδια πλευρά. Εδώ έχουμε πρόβλημα τώρα και η CR πάντα υποστηρίζει την επιστήμη. Εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτές τις αντιρρήσεις, γιατί α, κινούνται από κάποιους ιδεολογικούς φόβους. Η αξιολόγηση κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα είναι από τις πιο αυστηρές στον κόσμο και είναι αρκετά ασθεναρή για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα γενετικώς τροποποιημένα είναι όσο ασφαλή είναι και τα συμβατικώ καλλιεργούμενα προϊόντα. Ή ο κανονισμό για του γενετικού τροποποιημένου βεβαίω υποστηρίζεται από, τη, από, τα στατιστικά, από την επιστημονικά δεδομένα Τώρα βεβαίως εδώ παρεμβαίνουν και διάφορα πολιτικά θέματα, αλλά αν τα αφήσουμε αυτά να παρέμβουν θα ε, υποβαθμίσουμε την νομιμοποίηση όλου του συστήματος δείτε καταρχάς πώς μπορούμε να ε, κατακρίνουμε τους σκεπτικιστές για το κλίμα ή αυτούς που είναι αντίθετοι με τα εμβόλια που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, ενώ συστηματικά αγνοούμε τις, τα επαναλαμβανόμενα συμπεράσματα της ε, ΕΦΣΑ, τα οποία λένε ότι οι γενετικώς προποιημένοι οργανισμοί είναι απολύτως ασφαλείς. Κατανοώ βεβαίω, ότι κάποια από εσά έχετε πολιτικές αντιρρήσει, ε, καταναβαίνω τους χριστιανοδημοκράτε, που έχουν μια δική τους άποψη για το θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε το ότι παρόλο που ενώ μάλλον η, η χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών είναι περιορισμένη για κατανάλωση, Υπάρχει πολύ σημαντική χρήση για την παραγωγή και οι αντιρρήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και πλειοψηφία, μπορεί τελικώς να έχει πραγματικά καταστροφικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εμείς έχουμε επιφυλάξεις, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν έχω κανέναν άλλο να ζητά το λόγο. Ωραία. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Υγείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλια όλων. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλες τις παρεμβάσεις. Πρέπει να επιβεβαιώσω ότι όλα τα βήματα που έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει στα πλαίσια των ε, δικαιωμάτων της ε, εφαρμογής που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΦΣΑ έχει κάνει μια συνολική αξιολόγηση κινδύνου και έχει καταλήξει στο ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε διαβούλευση με την ΕΦΣΑ για το σχέδιο της νομοδότησης και όλα τα σχόλια έχουν ληφθεί υπόψη και από την ΕΦΣΑ. Επί τη βάση αυτή λοιπόν, επί τη βάση της θετικής νομοδότησης της ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις ε, προτάσεις της στην Επιτροπή. Και βεβαίως σωστά δεν παίρνουμε γνωμοδότηση από, την, από τις επιτροπές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η απουσία, η απουσία των ε, γνωμοδοτήσεων ή κομισιών θα πρέπει να, να μην μπορεί να ε, εγκρίνει. Πρέπει να, να καταλάβουμε ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και ο στόχος της, του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα γενετικώς τροποποιημένα που πάνε στην αγορά την Ευρωπαϊκή είναι ασφαλή. Λαμβάνοντας βεβαίω υπόψη και του παράγοντε που έχουν τονίσει κάποιοι από του παρεμβαίνοντε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αποφάσει για να επιβεβαιώσει κανεί την ασφάλεια επιμέρους μεμονωμένων προϊόντων δεν μπορούν να έχουν άμεση σύνδεση με τον όγκο των εισαγωγών από μία επιμέρους τρίτη χώρα ούτε με την επιτοχή των, επιτυχία, συγγνώμη, των ε, διεθνών δεσμεύσεων. Εδώ μιλούμε για την έγκριση επιμέρους μεμονωμένων προϊόντων για να εξασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλή. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της κλιματική ε, κλιματικής ε, αλλαγής ή της αποψήλωσης μέσω αυτού. Τούτου λεχθέντος η έγκριση αυτών των ιδιωτικοσωπημένων οργανισμών δεν υποβαθμίζει καθόλου την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων όπως εξήγησε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σήμερα το πρωί, για την πλήρη και συνεκτική στρατηγική. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι η έγκριση επιμέρους γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών δεν υποβαθμίζει σε κανένα βαθμό την συζήτηση που γίνεται για την ανάπτυξη πρωτεϊνούχων φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αν όντω είναι επιτυχής, θα διευκολύνει μειωμένη, την μειωμένη εξάρτηση από τι εισαγωγέ που έχουμε τώρα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο, παρα, ο, παρα, ο, ε, της παραγωγής εξαρτάται από τι πρωτεΐνες. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι πρωτεΐνες που εισάγονται είναι ασφαλείς. Αυτό είναι ο στόχο του κανονισμού τη νομοθεσία και έχουμε αυτή την εξάρτηση. Υπάρχει ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα προϊόντα προϊόντα. Ο στόχος λοιπόν όλης αυτής της συζήτηση για τα πρωτεϊνούχα φυτά δεν υποβεβάζεται από την έγκριση των ε, γενετικοσωπημένων οργανισμών. Αντίθετα, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, έτσι ώστε να μειωθεί η, ε, κατανάλωση αυτών των και η εξάρτησή μας από αυτές τις εισαγωγέ. Επίσης, η έγκριση των επιμέρους ε, γενετικοσωπημένων οργανισμών δεν, υποβαβεί, δεν υποβιβάζει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποψήλωση. Ποιος είναι ο στόχος να αυξηθεί η κατανάλωση ε, προϊόντων που δεν έχουν ε, υποστεί, ε, που δεν έχουν παραχθεί από, από ψηλωμένα δάση. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Το θέμα δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια όμως του γενετικοσωπημένου οργανισμού. Το θέμα είναι θέμα εξάρτησης και κατανάλωσης. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες για αυτό τους συγκεκριμένους γενετικοσωπημένους οργανισμούς που μπορούν να επιβαρύνουν την έγκριση. Γιατί αυτοί οι οργανισμοί είναι ασφαλείς. Η ΕΦΣΑ έχει συμπεράνει ότι είναι ασφαλής και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό για τους γαματαφόμικρων πρέπει να λάβει απόφαση και γι' αυτό πρέπει να είναι θετική απόφαση. Συμπερασματικά να πω ότι παρόλο που βεβαίω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτρέπεται, αν μπορώ να το πω έτσι, να αμφισβητήσει την, το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεπεράσει τις ε, εφαρμοστικές εξουσίες. Πρέπει να πω ότι έχουμε σεβαστεί τις ε, αρμοδιότητες που έχουμε, αλλά βεβαίως αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις και κάποιες αντιρρήσεις και βεβαίως ευχαρίστως να είμαστε σε διάλογο και να απαντήσουμε σε ό,τι χρειαστεί. Ελπίζω ότι η κατάληξη της συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχέδια ψηφίσματος ε, έχει καλύψει κάποιες από τις ανησυχίες και ελπίζω ότι θα διευκολύνει έναν καλό επικοδομητικό διάλογο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και να εφαρμόσουμε την νομοθεσία όπως έχει υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάποια χρόνια πριν. Σας ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η ψηφοφορία θα γίνει το απόγευμα και αν εγκριθούν οι αντιρρήσει, θα ξαναπισυφιστεί στην Ολομέλεια το θέμα στην επόμενη σύνοδο των Βρυξελών. Ε, και προχωρούμε ε, στο άλλο θέμα, στο επόμενο, που είναι Ε, το Παγκόσμιο Σύστημα Συλλογή Δεδομένων για την Κατανάλωση Μαζούτα από πλοία. Θα δώσω το λόγο τώρα ε, στην εισηγήτρια, την κυρία Γιούτα Πάουλου, και μετά στου σκιώδες εισηγητέ. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναθεώρησε την πρόταση η οποία ήδη έχει τεθεί σε ισχύ και έχουμε ε, συλλέξει και τα πρώτα δεδομένα για φέτος. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους τους παρόντες ότι η ναυτιλία είναι από τους λίγους κλάδους ε, εκτός από την ε, αεροπλοεία που δεν έχει καθόλου δεσμευτικούς στόχους και όποιος έχει διαβάσει το newsletter της Επιτροπής μας που βγήκε χτες θα είδε ότι αυξήθηκαν οι εκπομπές κατά 48% από το 90% από την αυτιλία ε, χωρίς να διαφαίνεται ε, μείωση. Μπορεί να αυξηθούν μέχρι και 200% μέχρι το 2050. Το σύστημα συλλογής δεδομένων μας είναι μεν καλό, ιδιαίτερα Ε, το σύστημα MRV που ελέγχει ε, το καύσιμο που μεταφέρεται. Πολύ καλό αυτό γιατί όλο και περισσότερο ε, ζητείται από το κλάδο να μετράει το αποτύπωμα άνθρακα Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το κάνει αν δεν ξέρει πόσο φορτίο μεταφέρει κάθε φορά το κάθε πλοίο. Ποιος είναι ο στόχος ε, να ε, συμμορφωθούμε με το σύστημα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, IMO, που έχει ένα σύστημα και λίγο διαφορετικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να μην υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια για τους πλειοκτήτες θα πρέπει να συμμορφωθούν, να, να συμπλησιάσουν το ένα σύστημα ε, το άλλο. Βέβαια, η συλλογή δεδομένων δεν ταυτίζεται με τη μείωση των εκπομπών, έτσι και όποιος διάβασε χτες τα νέα είδε ότι 11.000 επιστήμονες καλούν σε άμεση δράση για την κλιματική αλλαγή. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τώρα σημαντικά βήματα. Και κατά την άποψή μου το πρώτο είναι να ακολουθήσουμε την έκκληση της κυρίας Φόντερ Λάιεν και να συμπελάβουμε και την αυτιλία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και να έχει το μερίδιο που της αναλογεί. Και το 20% των εσόδων μπορούν να διοχετευθούν για καλύτερους κινητήρες, καλύτερα πλοία που να ρηπαίνουν λιγότερο και τελικά να βρούμε και πιο δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπέ της ναυτιλίας. Αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Θα πρέπει όμως να θεσπιστεί αν δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε το σύνολο των κλιματικών μας στόχων. Ε, με μεγάλη χαρά περιμένω να ακούσω τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι άλλοι συνάδελφοι, οι σκιώδεις συζητητές. Ευχαριστώ πολύ ωραία μετάβαση. Θα περάσουμε μέσω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην παρουσίασή της και μετά θα ακούσουμε τους σκιώδεις ηγητές. Θα παρακαλέσω την κυρία Μπεατρίξ Ιόντι από τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, χαρά μας που είμαστε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο για να σας εξηγήσουμε ποια είναι η πρόταση αυτή που αποκαλούμε MRE για την παρακολούθηση. Ε, μισό λεπτό τώρα να ξεκινήσω και τις διαφάνειες. Ε, όπως είπε μόλις η Γιούτα Πάουλους, ε, είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας με συνολικό, το συνολικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό και θα σας αναφέρω λοιπόν όλα αυτά που περιλαμβάνονται και σε αυτήν την πρώτη διαφάνεια. Το πλαίσιο ποιο είναι λοιπόν. Έχουμε έναν ε, τομέα κλειδί που μεταφέρει 80% του παγκοσμίου εμπορίου. Είναι η ναυσιπλοεία. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Μιλάμε για 2 με 3% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ψηλότερα σε εκπομπές δηλαδή από οποιοδήποτε κράτος μέλος από μόνο του. Αν ήταν μια χώρα, η ναυσιπλοή θα ήταν υπαριθμόν 6 ε, στις εκπομπές. Αναμένεται να αυξηθεί και μάλιστα υπάρχουν διάφορα σενάρια που συνδέονται με τα εμπορικά σενάρια που είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν, αλλά όλοι συμφωνούν ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση των εκπομπών οι Ευρωπαίοι πλειοκτήτες ε, ελέγχουν το 1 τρίτο του παγκοσμίου εμπορικού στόλου. Πολύ μεγάλος ε, τομέας λοιπόν με δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομική αξία βέβαια. Να σας δείξω σε ένα πιο όμορφο σχέδιο ε, γράφημα τα νούμερα που μόλις σας ανέφερα. Μιλάμε για 36% του συνόλου του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου και για το εξωτερικό εμπόριο καλύπτει η ναυσιπλοεία το 75% και όπως σας είπα προηγουμένως το 80% ε, αφορούσε παγκόσμια νούμερα. Τώρα, ποιο είναι το πλαίσιο. Χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις επιγόντως. Ε, ο διεθνής τομέας της ναυσιπλοής είναι ο μόνος που δεν περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όλοι οι τομεί, όπως είπε και η νέα πρόεδρος και δήλωσε, όλοι οι τομεί και η ναυσιπλοεία θα πρέπει να συμβάλλουν στην ε, επίτευξη των στόχων τη συμφωνία του Παρισιού. Να επαναλάβω το τρίτο σημείο, το οποίο είναι πολύ προσφυλές στο Κοινοβούλιο και Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας ε, Εκπομπών που καλεί σε δράση σε επίπεδο ΑΕΜΟ, δηλαδή Διεθνούς Οργανισμού ε, Ναυσιπλοείας και να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από το 2023. Βεβαίω σε διεθνέ επίπεδο, το διεθνέ επίπεδο είναι αυτό που πρέπει να ενθαρρυνθεί διότι πρόκειται για διεθνή αγορά και εργαζόμαστε επ' αυτού και τώρα θα επανέλθω, μάλλον θα έλθω στην μέτρηση γιατί δεν είναι η ε, παντού ακόμα και αν η μέτρηση ήδη οδηγεί σε κάποιο κομμάτι μείωση των εκπομπών. Λοιπόν, τώρα να μην σας ε, κουράσω με όλα τα ακρονίμια του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλία για τον δίκτυο, ας πούμε, ενεργειακής απόδοσης ή για την διαχείριση των πλοίων. Αυτοί που δουλεύουν στην αυσιπλοεία γνωρίζουν όλα αυτά, αλλά να σας πω γενικά Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ξεκινήσε το 2011 με την νομοθεσία για την ε, επάρκεια σε ενέργεια, την απόδοση μάλλον σε ενέργεια, όχι πολύ αποτελεσματική. Ε, μετά υπάρχει το σύστημα συλλογής στοιχείων του IMO. Ας ξεχνάμε ότι προήλθε αυτό από ευρωπαϊκό σύστημα δεδομένων. Αρχικά ήταν ευρωπαϊκό σύστημα και μετά ο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλία το χρησιμοποίησε. Μετά, το 2018, πολύ σημαντική ημερομηνία, γιατί ε, ο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλία όρισε στόχου μείωση, τουλάχιστον 50% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τις τιμέ του 2008 και όσο είναι δυνατόν, όσο γίνεται πιο σύντομα, να ε, μειωθεί η ένταση χρήσης άνθρακα. Τώρα λοιπόν, τι έχουμε από ρυθμιστική άποψη. Έχουμε επιτάπητο, είναι στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προ συζήτηση αυτό ο κανονισμό ε, του 2015. Να σα θυμίσω ότι ήταν ένα πρώτο καλό βήμα στην συλλογή και επαλήθευση εκπομπών και στοιχείων. Δεν ήταν συλλογή στοιχείων στο δικό μου καιρό να επαέλθει διαφάνεια ώστε να υπάρχει επιλογή και να αλλάξουν και οι συμπεριφορές και να ενημερωθούμε για τις μελλοντικέ αποφάσεις. Στη συνύπαρξη των δύο συστημάτων. Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα από το 2015 και έχουμε το σύστημα του IMO από το 2016 και έχουμε μια ρήτρα στην MRV, το άρθρο 22.3, που ορίζει ότι σε περίπτωση διεθνούς συμφωνίας για παγκόσμια παρακολούθηση θα προσαρμόσουμε και θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Τώρα αντιμετωπίζουμε την, τον κανονισμό IMO περί στοιχείων. Τώρα, έχουμε αρμονική εκπροσώπηση και ε, ε, ε, εφαρμογή και θα εστιάσω στο δεύτερο σημείο, δηλαδή την διαφάνεια ώστε να εφαρμοστεί αυτή η Από τον Ιούλιο φέτος έχουμε από 11.600 σκάφη που ε, ε, πιάνουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Έχουμε τώρα αξιολόγηση αντικτύπου, έχουμε την πρώτη επιλογή ε, που βασίστηκε στις προηγούμενες αξιολογήσεις αντικτύπου όπως σας είπα, δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν, ήταν ένα κάποιο δεύτερο βήμα. Έχουμε λοιπόν τον πρώτη επιλογή του να μείνει έτσι ως έχει η νομοθεσία. Δεύτερον, να διατηρήσουμε τις βασικές μας αρχές. Και τρίτη επιλογή είναι η σύγκληση, δηλαδή πλήρης ε, εναρμόνιση με τον ε, IMO. Λοιπόν, έχουμε το θέμα της διακυβέρνησης που είναι σημαντικό γιατί εξετάζουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση γιατί σημαίνει ότι ε, ένα σκάφος το οποίο ταξιδεύει από το Ρότερνταμ στην ε, ε, Μασαλία δεν θα αναφερθεί ένα κινέζικο σκάφος Γι' αυτό και οι δύο αυτές επιλογές ε, απορρίφθηκαν. Σύγκριση των επιλογών τώρα. Θα, εδώ θα προχωρήσω πιο σύντομα. Η, η μέση οδός ήταν αυτή που προτιμήθηκε, η παριθμό 2. Η τρίτη δεν ε, υπήρχε περίπτωση η, η διαφάνεια να μην παρακολουθείτε. Είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε ευρωπαϊκό σύστημα ε, εποπτείας το ένα, το να μην κάνουμε τίποτα και να αφήσουμε ε, το βάρος της, ε, των εκθέσεων. Αυτό, ούτε και αυτό ήταν ικανοποιητικό και γι' αυτό ακολουθήσαμε την δεύτερη οδό. Ποια είναι τα βασικά ε, σημεία αυτής της πρότασης. Πρώτον, έχουμε την υποχρέωση της, ε, της εταιρεία να αναφέρει εάν αλλάξει εταιρεία τι θα συμβεί. Η θελοντική αναφορά του φορτίου που μεταφέρεται, αυτό ήταν σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Να θυμίσω πως ο ΑΕΜΟ δεν περιλαμβάνει αυτό το θέμα, αυτό δηλαδή το φορτίο που μεταφέρεται. είναι σημαντικό το, το βάρος, το ο φόρτος. Γι' αυτό το είπαμε ότι θα γίνεται αυτό εθελοντικά. Το άλλο κομμάτι είναι η συγγήτρια, όπως ανέφερε, έχουμε κορεπέρ τη Δευτέρα, ε, μάλλον, συγγνώμη, έχουμε εντολή της κορεπέρ από την περασμένη εβδομάδα. Να σας πω τώρα ποια είναι τα καλά νέα για την ε, ε, υπάρχουσα εποπτεία. Για πρώτη φορά έχουμε στοιχεία για τις εκπομπές από 11.600 σκάφη τα οποία πιάνουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια εκπροσωπούν 139 εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και από του χρόνου θα κάνουμε τη δική μας καταμέτρηση και έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για εντυπωσιακό κύκλο, πρώτο κύκλο συμμόρφωσης η Κομισιόν ήδη τα έχει δημοσιεύσει στην Μαρβή τη βάση δεδομένων που φιλοξενεί το MRV. Ε, ε, ε, Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να δημοσιεύονται και να είναι διαθέσιμα στο κοινό. Και τον Ιούλιο θα κάνουμε και την ε, αξιολάγηση. Αυτό είναι μια πρώτη γεύση. Και στην επόμενη έκθεση θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Και είναι τώρα η κατάσταση πρόοδου. Όπως σας είπα, το σύστημα MRV λειτουργεί, αποδίδει, είναι πολύ σημαντικό πολιτικής άποψης να αξιολογήσουμε το θέμα των εκπομπών στον τομέα της ναυτιλίας. Εάν δεν μπορέσουμε να... θα πρέπει να συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα για παρακολούθηση. Είναι ένα πρώτο βήμα για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο ή στρατηγική. Και γι' αυτό και έχουμε μια μερική προσαρμογή και ευθυγράμμιση και με το σύστημα του Θα Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους Ισκιώδης και μετά στην εισηγήτρια πάλι στο τέλος της συζήτησης βέβαια. Αλλά και στην Κομισιόν θα ξαναδώσω το λόγο εάν σας απευθυνθούν ερωτήσεις. Αρχίζουμε λοιπόν με το ΕΛ και τον Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τυπικά κάνουμε συζήτηση για δεδομένα τα οποία συλλέγουμε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για τις εκπομπές ε, της ναυτιλίας που βλάπτουν το περιβάλλον και το κλίμα. Βεβαίως, θα πρέπει με μεγάλη λεπτομέρεια να συζητήσουμε την νομοθεσία, να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά επίσης, είναι προφανές ότι τίθεται το ερώτημα τι θα τα κάνουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε. Άντε, συλλέγουμε δεδομένα, δεν θα πρέπει να έχουμε και κάποιες ε, συνέπειες. Αλλιώς δεν είναι πραγματικά ικανοποιητική η κατάσταση. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν εξήγηλε στην ομιλία της ότι θα ε, είναι απαραίτητη και αναγκαία συμμετοχή της ναυτιλίας στην αντιμετώπιση αυτών των στόχων του περιβάλλοντος. Και θα πρέπει να αποφανθούμε και να αξιοποιήσουμε την έκθεση της κυρίας Πάουλους για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Από τη μια έχουμε το θέμα αυτό προφανώς και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ότι ανατόνο και κατά ε, η ναυτιλία είναι πιο φιλική προς το κλίμα σε σχέση με την αεροπλοεία ή με την κυκλοφορία την οδική στους αυτοκινητοδρόμους. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν να μην αποφασίσουμε μέτρα που να ανατρέπει την κατάσταση, δηλαδή να υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση για την αυτιλία. Επίσης έχουμε το θέμα, όπως πάντα, της ανταγωνιστικότητας και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία δεν θα βλάψουν την Ευρώπη. Εδώ πρόκειται για όλα τα πλοία τα οποία ελιμενίζονται ε, στα ευρωπαϊκά λιμάνια και όχι μόνο για ε, τα ε, πλοία που έχουν συγκεκριμένη σημαία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε 250% αύξηση των εκπομπών και μείωση εκπομπών είναι σχετικά περιορισμένη ως προς το κόστος. Ε, και αυτό είναι και δίκαιο απέναντι σε άλλες ε, μορφές και μέσα μεταφοράς που επιβαρύνονται. Το είπε και η Ursula von der Και στην παρουσίαση εδώ είδαμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ, η κοινή γνώμη. Η ναυτιλία είναι ένα θέμα στο οποίο ο κόσμος περιμένει να αντιδράσουμε για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Άρα δεν θα πρέπει να μας απασχολούν και να συζητούμε μόνο τα τεχνικά ζητήματα, αλλά να στείλουμε και ένα πολιτικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα συμπεριληφθεί η ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πώς το φανταζόμαστε για να μην βλάψει τον ανταγωνισμό, για να μην το παρακάνουμε, αλλά ότι πρέπει να ασχοληθούμε και ασχολούμαστε με το θέμα, νομίζω ότι έχει νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σοσιαλιστέ και δημοκράτε η κυρία Γιώτελαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Γιώργη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε και μας έκανε σήμερα την παρουσίαση. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την αυτιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αυξηθούν κατά 86% ε, σε σχέση με το έτος αναφοράς του 1990. Μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε δε από την εισηγήτρια αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως έχουν τα παγκόσμια στοιχεία και μέχρι το 2050 αναμένεται αύξηση μέχρι και 200%. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Βρισκόμαστε μεσούσεις μιας έκτακτης ανάγκης για το κλίμα οι πάντες ε, σε όλους τους τομείς και όλη η κοινωνία πρέπει να μετασχηματιστεί και να ευθυγραμμιστούμε με τους στόχους της Συμφωνίας ε, του Παρίσιου. Ένας από τους ε, τομείς αυτούς που εξαιρούνται περιέργως είναι η ναυτιλία, γιατί πλέει κάτω από τα ραντάρ εδώ βλέπουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο κόσμος έχει επαναστατήσει. Βλέπουμε ανθρώπους σε τα λιμάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βλέπουν αυτά τα μεγάλα πλοία ε, ε, τα οποία είναι ελιμενισμένα και παρόλα αυτά ε, έχουν αναμένους τους κινητήρες και ρηπαίνουν πάρα πολύ. Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο το κλίμα, αλλά και την υγεία των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, συμφωνώ με τον Πέτερ Λίζε. Ως νομοθέτες θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα τώρα να σταματήσει να είναι λαθρεπιβάτης η ναυτιλία όταν οι πάντες ε, αυξάνουν τις προσπάθειες. Ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουμε δείξει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Χρειάζεται εναρμόνιση και ευθυγράμμιση της δικής μας νομοθεσίας με τους κανόνες του IMO. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα ρίξουμε εμείς τα δικά μας πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο. Ε, χρειάζεται παγκοσμίω να αυξηθεί η προσπάθεια. Και εδώ υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να βελτιώσουμε στην πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής. Κυρία Γιώργη, γνωριζόμαστε από χρόνια με το ETS, το σύστημα εμπορίας εκπομπών και ήδη από τότε ξέρατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ πιο φιλόδοξο και θέλαμε και η ναυτιλία να μειώσει ε, ε, τις εκπομπές. Ζητήσαμε νομοθεσία από παλαιότερα. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει όχι, αλλά να χρησιμοποιήσουμε το MRV, το σύστημα παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα το κάνετε αυτό για τη μείωση των εκπομπών. Ε, με χαρά θέλω να σας ακούσω τώρα, να μας απαντήσετε, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Εμείς στο Κοινοβούλιο ε, πρόκειται να αρχίσουμε την νομοθετική μας ε, δράση για αυτή την πρότασή σας και πώς βλέπετε να συνδέεται το MRV με την εισαγωγή συγκεκριμένων στόχων μείωσης εκπομπών για ε, τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει έρθει η ώρα και με τα στοιχεία που συλλέγονται από το MRV θα μπορούσαμε να έχουμε μία πρόταση για να μειωθούν οι εκπομπές της ναυτιλίας οι βλαβερές για το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο, Πρόεδρος. Από την ομάδα Ρινιού, η κυρία Κατρίν Σαμπού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, μια διαπίστωση. Εδώ και χρόνια ο κλάδος κινητοποιείται για να μειώσει τις εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου και μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό το σύστημα του MRV είναι πάρα πολύ τεχνικό και έρχεται εδώ στο Κοινοβούλιο προς ενώ νέες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για το κλίμα δημοσιεύονται και μας λέουν ότι από τους δύο βαθμούς θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, να μιλήσουμε για 1,5 βαθμό Κελσίου αύξησης της θερμοκρασίας. Και βλέπετε πόσο απέχει η νομοθεσία στη σύλληψη της και στην υιοθέτησή της από την εφαρμογή. Θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι στην Ευρώπη, μεν, βεβαίως, να λαμβάνετε υπόψη και να συνυπολογίζετε και το φορτίο και η διαφάνεια των δεδομένων, αλλά πρέπει να φτάνουμε και στους στόχους. Ο στόχος ποιος είναι. Να δούμε ποια είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα των σκαφών. Εγώ συμφωνώ με την απλούστευση, ε, τη διοικητική, αλλά δεν θα πρέπει τώρα αυτό να συνιστά οπισθοδρόμηση σε σχέση με τις φιλοδοξίες και την έκτακτη ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές της ναυτιλίας. Ε, εγώ έχω 90% και όχι 80% του εμπορίου ε, ε, που γίνεται με την αυτιλία. Βεβαίω, υπάρχει σύστημα εμπορία εκπομπών και ανταλλαγή εκπομπών. Δεν διαφωνώ να μπει στο ETS η ναυτιλία βεβαίω. Αλλά προσοχή. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι μια λύση που θα σπρώξει κάποιους πλειοκτήτες προς τα λεγόμενα πράσινα σκάφη, green ship. Γιατί υπάρχουν κάποιοι πλειοκτήτες, ιδιαίτερα οι Γάλλοι εφοπλιστές, ε, που θέλουν να βελτιώσουν τα σκάφη τους ε, και προσοχή να μην το παρακάνουμε. Γίνεται λόγος για εκπομπές, αλλά δεν είναι μόνο εκπομπές, είναι και η βιοπικιλότητα ε, των θαλασσίων ειδών. Έχω πρόβλημα εγώ ε, για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ε, το χρόνο ναυσιπλοείας. Τι θα πει πότε είναι εμπλό και πότε δεν είναι εμπλό. Ακόμα και λιμενισμένο να είναι το σκάφος, αν δεν παίρνει ρεύμα ε, από τον προβλήτα, οι κινητήρες είναι σε λειτουργία. Γιατί και εγώ ε, έχω σκάφος και ξέρω Ας πούμε, στην ε, Μαρσαλή αυτή τη στιγμή, στο λιμάνι, ε, κάνουν διαβήματα οι πλειοκτήτες έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροδότησης του σκάφους από τη στεριά για να σβήνουν τους κινητήρες. Υπάρχουν πολλά θέματα ε, ε, που μπορούμε να συζητήσουμε, όπως είναι η μείωση της ταχύτητας, ας πούμε, των σκαφών. Ορισμένοι πλειοκτήτες το έχουν αυτό ε, σκεφτεί ε, και θα μπορούσαμε και εμείς να το σκεφτούμε. Γιατί μπορούν έτσι να μειωθούν πολλοί εκπομπές και να προωθήσουμε και τα green ships. Δηλαδή υπάρχουν Τώρα, συστήματα υβριδικά, ε, αντί τη, ε, τη θερμοκίνηση να υπάρχει και μια ε, κίνηση με την αιωλική ενέργεια, ας πούμε ένα 30%. Εγώ εδώ και καιρό θέλω η Ευρώπη να έχει μια βιομηχανία ανακύκλωσης των σκαφών και να μην τα στέλνουμε στην άλλη άκρη της γης για να ανακυκλωθούν τα παροπλισμένα. Επίσης, ε, δεν θέλω να έχουμε μόνο ένα green deal, αλλά και ένα blue deal, ε, μια γαλάζια πράσινη συμφωνία δηλαδή, για να μην εξαιρείται η ναυτιλία από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ζωέλ ε, Μελά από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Απουσιάζει. Η κυρία Μανά, δεν υπάρχει κανείς από το ID. Ωραία. Από το ICA. E Ο κύριος Βόντρα, παρακαλώ. Well, thank you. I I... Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι συγκεκριμένο. Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως σε κάθε τομέα την, την ε, κλιματική αλλαγή αν είμαστε όντως πεπισμένοι ότι είναι ένα θέμα παγκόσμιο, άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Άρα λογικό είναι να συμπεριλάβουμε και την αυτιλία στα μέτρα που θα λάβουμε. Λογικό. Ακούγεται, δεν έχω να προσθέσω κάτι σε όλα όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Γκουέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπίσει το υπάρχον σύστημα MRV για τη συλλογή δεδομένων σε σχέση με τις αδυναμίες που έχει το σύστημα του IMO για τη συλλογή δεδομένων. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το, το, το, το σύστημα του, του IMO δεν είναι τόσο διαφανές όσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα δεν δημοσιεύονται, τα, τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν εξ, επαληθεύονται ανεξάρτητα από ένα τρίτο ε, μέρος και αυτά τα στοιχεία ε, ε διαφάνειας στο, που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα έχουν ε, επιβιώσει και στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύστημα συλλέγει στοιχεία για το τονάζ και όχι για το φορτίο που ε, κουβαλεί το πλοίο. Και το υπάρχον σύστημα και ο σχετικό κανονισμό MRV ζητά να, τα, τα πλοία να στείλουν δεδομένα για το φορτίο που μεταφέρουν για την ε, ε, ενεργειακή απόδοση. Το μεταφερόμενο φορτίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δούμε τις εκπομπές σε σχέση με το φορτίο του και να δούμε την ε, επάρκεια σε σχέση με τον άνθρακα. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε διαφορά μεταξύ ενός άδειου πλοίου και ενός πλοίου με φορτίο. Έχει υπολογιστεί ότι ένα τρίτο των πλοίων που έρχονται στα ευρωπαϊκά λιμάνια δεν κουβαλούν τίποτα άλλο πέραν των καυσίμων τους. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε γιατί το σύστημα του ε, IMO είναι τόσο μυστικοπαθές. Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα του IMO ε, ελέγχεται από τους ε, εφοπλιστές και από τα διάφορα κράτη. Η, προ, η πρόταση Κομισιόν που επιβάλλει πίεση ώστε να συλλέγονται τα στοιχεία και για το φορτίο είναι σημαντική. Αλλά δεν έχει, δεν κάνει, δεν έχει καμία σημασία τελικώς για τους εφοπλιστές. Τα κράτη ε, όπως ε, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία ε, χρησιμοποιούν το σύστημα MRV σε, σχέση με το, σε αντίθεση με το πιο αδύναμο του IMO, αλλά και το σύστημα MRV της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βελτιωθεί. Ο κανονισμός ζητά υποβολή εκθέσεων μόνο για τις εκπομπές διοξιδίου του, άνθρακα, του άνθρακα, αλλά θα πρέπει να, το, να το χρησιμοποιήσουμε και για εκπομπές άλλου είδους, μεθανίου. προς το παρόν, Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και με το project για το υγροποιημένο αέριο στην ε, Ιρλανδία. Με φορτία που έρχονται από την Αμερική. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο οι εκπομπές λαμβάνονται υπόψη. Μάλλον είναι λίγο ανόητο αυτό το σύστημα. Επίσης, τα, συστήματα, τα στοιχεία που δημοσιεύονται δημοσιεύονται μόνο για τις εκπομπές αναπλή, αλλά όχι εταιρεία. Αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο, γιατί συνήθως για το, για το σύστημα MRV ε, το αντίθετο ισχύει. Γιατί λοιπόν αποκρύπτονται αυτές τις πληροφορίες. Αν ε, ψάξω στο Google το όνομα ενό ε, πλοίου, μπορώ να βρω και τον ιδιοκτήτη του. Αλλά είναι αδύνατο να δω ποιε είναι οι εκπομπέ μια εταιρεία που έχει έναν αριθμό σκαφών και πρέπει να κάτσω να ψάξω ας πούμε μια, τις 1100 σελίδες μιας έκθεσης για να το βρω. Είναι αδύνατο λοιπόν να γίνει αυτό για όλα τα πλοία, κυρίως επειδή πολλές είναι από, πολλά, ε, είναι από εταιρείες ε, που, είναι, που έχουν μόνο μια ταχυδρομική θηρίδα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε γενικώ την ε, συνολική εικόνα για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα ανά εταιρεία. Και πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε περίπτωση που έχουμε μόνο ένα ταξίδι, μόνο χρήση του πλοίου για ένα μήνα, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι operators είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να πληρώσουν το τίμημα των εκπομπών και να τηρούν τα πρότυπα για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες σχετικά και νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο απλό να είναι ο υπεύθυνο ο, ο ιδιοκτήτη του πλοίου. Είναι πολύ πιο απλό. Μέχρι στιγμή το σύστημα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε και θα υποβάλουμε τροποποιήσεις για μέτρα μείωση ε, και για, τα, για, τις, για μηδενικέ ε, εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα και συνολικά για μηδενικέ εκπομπέ. Ευχαριστώ. Ωραία. Να περάσουμε στο Catch the Eye τώρα. Από το ΕΛΚ πρώτα. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι από, το, από την περήφανη Δανία και χαίρομαι που μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί είναι σημαντικό, όπως είπε και ο τελευταίος συνάδελφος, ότι πρέπει να ενισχύσουμε το MRV, το σύστημα ως εργαλείο για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η ναυτιλία ε, ε, επιδρά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχω ένα ερώτημα, ωστόσο. Αν το κάνουμε αυτό συμπεριλαμβάνοντας την ναυτιλία στο ETS, στο σύστημα ανταλλαγής εκπομπών, αν θέλουμε να βελτιώσουμε σε διεθνές επίπεδο την ναυτιλία και πώς μπορεί αυτή να πρασινίσει ως το δυνατόν περισσότερο. Ίσως να πρέπει να σχεδιάσουμε ένα διαφορετικό εργαλείο για τη μέτρηση. Για να υποστηρίξουμε το MRV και για να δείξουμε ότι οι ευρωπαϊκές πλειοκτήτριες εταιρείε είναι έξι φορές λιγότερο επιθετικές προς το περιβάλλον σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες παγκοσμίω. Οπότε ρωτώ, μπορούμε να είμαστε ήδη από τώρα σίγουροι ότι μέσω του ETS είναι ο καλύτερος δρόμος για να αλλάξουμε την βιομηχανία της ναυτιλίας και να την καταστήσουμε πιο πράσινη. Ίσως ένα άλλο εργαλείο που θα μπορούσε να κάνει την, το σύστημα πιο προσαρμόσιμο ε, εντός του IMO να χρειάζεται σε αυτή τη φάση. Γιατί πρέπει να σεβαστούμε ότι και το σύστημα ETS δεν κάνει αυτό που πρέπει. Αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε. Και εκεί υπάρχει μια αναδιάρθρωση ή χρειάζεται μια αναδιάρθρωση. Οπότε αν θέλουμε όντως να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή ε, Ναυτιλία και το κλίμα, ίσως να πρέπει να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί στην προσέγγιση και στην σχεδιασμό του εργαλείου που θα έχουμε. Και επίσης το ρωτώ αυτό, γιατί υπάρχει και το θέμα των ε, υποχρεώσεων ή το κατά πόσο είναι επιλογή να έχουμε πληροφορίες για το μεταφερόμενο φορτίο. Αυτό το είναι ε, υποχρεωτικό, δεν θα είναι επικουρικό, δεν είναι ε, επιλογή. Είναι σημαντικέ οι πληροφορίε αυτέ. Οπότε είναι περίεργη και η λογική πίσω από αυτέ τι συστάσει τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί προτείνει η Κομισιόν να είναι προαιρετικό δηλαδή. Θέλουμε ούτω ή άλλω έναν πράσινο δρόμο για την ναυτιλία. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά όμω ακόμα και χαίρομαι πολύ που μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την κύριο Κόκαλη, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ από μικρό περήφανο ναυτικό κράτος είμαι. Και ε, θα ήθελα να σας πω... IMO είναι ε, οργανισμός των ε, Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι του κλάδου ιδιωτικός φορέας. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και παίρνονται διεθνείς αποφάσεις εκεί. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Συγγνώμη, κύριε Γουόλας, έχετε αναμένο το μικρόφωνο σας και δεν βλέπουμε τον κύριο Κόκαλη. Έλεγα λοιπόν ότι δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι η ναυτιλία ε, θα πρέπει να ρυθμιστεί όπως και κάθε κλάδος που εκπέμπει η διοξίδιο του άνθρακα. Δυστυχώς στη Συμφωνία των Παρισίων ε, τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν μια αναβολή 5 ετών. Ωστόσο, έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα ε, για την αυτιλία να ρυθμίζεται παγκοσμίω παρά σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορα συστήματα ρύθμισης, το ETS, η διαρροή του άνθρακα και όλα αυτά ε, πώς να το πω, χρειάζεται μεγαλύτερη μελέτη πριν ε, προβούμε σε οποιαδήποτε δράση. Και το γεγονός ότι η IMO προτείνει ένα σύστημα αντίστοιχο με το MRV έχει σημασία. Ωστόσο, το δικό μας MRV είναι πολύ καλύτερο από εκείνο του IMO και η λύση εδώ είναι να οθήσουμε το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας να υιοθετήσει το δικό μας MRV, το οποίο φυσικά καταγράφει όλα τα ε, θέματα φορτίου, τρίτες χώρες, ε, και τα λοιπά, ε, πολύ σημαντικά δεδομένα που πρέπει να είναι και δημόσια. Ένα τελευταίο. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να τα δούμε διαφορετικά, ξεχωριστά. Άλλο τα λιμάνια, άλλο τα πλοία. Τα λιμάνια είναι πολύ προβληματικά ως προς τον ατμοσφαιρικό αέρα που υπάρχει εκεί για τους κατοίκους της ε, στεριάς. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα ε, ε, το να ε, είναι τα πλοία στο λιμάνι δεν μπορούν να σβήσουν τους κινητήρες γιατί δεν θα έχουν ρεύμα. Άρα χρειάζεται ηλεκτροδότηση από το λιμένα. ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Θα δώσω και πάλι το λόγο στην εισηγήτρια και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη. Νόμιζα ότι αντίστροφα γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Πρόεδρος, δεν ξέρω, αν έχετε ερωτήσεις... Αν έχετε ερωτήσεις, σας δίνω το λόγο. Θέλετε να ακούσετε πρώτα τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά να μιλήσετε εσείς. Ναι, ναι, πολύ θα με ενδιαφέρει να ακούσω την Κομισιόν και να μετά να κλείσω. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ε, ωραία. Απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και πάρα πολύ εύστοχες. Ε, θέλω να επανέλθω στα διαδικαστικά. Αυτή η αναθεώρηση που έχουμε σήμερα επιτάπητος ε, είναι ε, η αναθεώρηση του σύστηματος MRV, που είναι ένα σύστημα παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης στο 22-3. Εγώ ε, αισθάνομαι έτσι πως σας τα λέω σαν καλή γραφειοκράτης, αλλά είναι καθήκον μου να σας φέρω το θεσμικό πλαίσιο. Σε αυτόν τον κανονισμό τι ορίζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποχρεούται να κάνει κάποια πράγματα και με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις. Εμείς σε αυτό περιοριζόμαστε αυστηρά. Ε, στις αλλαγές που προτείνονται έτσι ώστε να εφηγραμμιστεί έστω και μερικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ε, IMO. Κατά την άποψή μας οποιαδήποτε αλλαγή ε, σε αυτόν τον κανονισμό θα άλλαζε το πεδίο εφαρμογής, το ETS και τα άλλα μέτρα. Όλα αυτά μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού. Όπως γνωρίζετε, δεν είναι η συζήτηση συνολικά για ε, το ETS. Ε, ξέρω πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος της ναυτιλίας για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι. Και ε, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που μας έχει δώσει η εκλεγμένη πρόεδρος, θα γίνει μια μελέτη αντικτύπου και μετά εν ευθέτω χρόνο θα υποβληθεί και νομοθετική πρόταση. Αλλά τονίζω, για να γίνει αυτό χρειάζεται πλήρης μελέτη αντικτύπου και ανάλυση των διαφόρων ε, δράσεων που έχουμε, επιβολή τέλους, ETS και θα πρέπει να γίνει και διαβούλευση με τον κλάδο. Ε, υπάρχει παρελθούσα εμπειρία, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το ιδεώδες ε, να βασιστούμε σε αυτή. Θα πρέπει να γίνει νέα διαβούλευση και νέα εκτίμηση. Θεωρεί αυτό σημαντικό και η κυρία Φόντερ Λάιεν θέλουμε εν ευθέτω χρόνο να έχουμε δράση και για την αυτιλία, αλλά πρώτα να γίνει σωστή διαβούλευση, καλή ανάλυση και καλύτερη νομοθεσία. Αυτά ε, για τα όσα είπαν ο κύριος Λίζ, η κυρία Γιούτελαντ, η κυρία Σαμπό, η κυρία Βάις, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Γουόλας. Να έρθω ε, στο φορτίο λίγο ε, και να διευκρινίσω. Ο IMO δεν ε, ε, έχει υποχρέωση αναφοράς του φορτίου. Ε, μιλούν για χωρητικότητα καινού φορτίου, dead weight donuts. Εμείς μιλούμε για εθελοντική αναφορά του φορτίου. Για ποιο λόγο? Για δύο λόγους. Πρώτον, στη διαβούλευση ήταν ξεκάθαρο το αίτημα ότι το να είναι εθελοντικό γιατί θα αυξηθεί η γραφειοκρατία και το δεύτερο είναι ότι δεν διακυβεύει το στόχο της αλλαγής συμπεριφοράς και ε, γιατί υπάρχουν οι άλλες παράμετροι για την ενεργειακή απόδοση που μας δίνουν ε, αρκετά χρήσιμα στοιχεία και επαρκή. Βέβαια να γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε ενημέρωση για το φορτίο ε, μπορούμε να υπολογίσουμε καλύτερα το αποτύπωμα άνθρακα ε, και έχει δείξει ενδιαφέρον ε, ένα τμήμα του κλάδου στο να συνεχίσει να συλλέγει αυτή τη σημαντική πληροφορία. Ένα άλλο σημαντικό που είπε η κυρία Σαμπό γιατί το διοξίδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων στους λιμένες. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στην πρότασή μας. Η τελευταία ερώτηση είναι η δράση Spirit. Είναι ιδιαίτερα προσφυλής και στον κλάδο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε, έχουμε μια σημαντική ε, διάσκεψη στο Λονδίνο την άλλη εβδομάδα, στον IMO. Εμείς υποστηρίζουμε τα μέτρα Ε, α, για την ταχύτητα, συγγνώμη, την ταχύτητα, για τη μείωση της ταχύτητας ε, των σκαφών. Ε, γιατί έτσι θα μειωθεί και η εκπομπή διοξιδίου άνθρακα. Back to the rapporteur to end this debate. Thank you and thanks for all for their contribution. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για, την... για τις παρεμβάσεις να απαντήσω σε αυτή την τελευταία μου παρέμβαση. Κύριε Λίζε, βεβαίως πρέπει να μην, υπάρχουν, ε, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση στα μέτρα που θα λάβουμε. Ε, εννοείται αυτό. Δεν πρόκειται να επιβάλλουμε μέτρα μόνο σε κάποιους εφοπλιστές. Όλοι θα πρέπει να τηρούν τα ίδια μέτρα, τους ίδιους κανόνες. Και χαίρομαι που πολλοί από εσά ε, θέσατε το θέμα της μείωσης των ε, εκπομπών και όχι της αντιστάθμισης αυτών. Απογοητεύτηκα βέβαια λίγο που λέει η Κομισιόν ότι ναι, αλλά στο MRV υποχρεούμεθα να ε, κάνουμε καταγραφή, γιατί το MRV ε, είναι το πρώτο βήμα και στα εισιτηλικές σκέψεις μιλάει για μείωση εκπομπών. Πάνω από 11 χρόνια πριν είχαμε μια οικονομική κρίση στην ε, Ευρώπη που ξεκίνησε και είχαμε ε, καθορίσει κανόνες και για να διασφαλίσουμε το οικονομικό μας σύστημα. Γιατί δεν μπορούμε να σώσουμε το ε, κλιματικό μας σύστημα αντιστοίχως. Το θέμα δεν είναι να ξεπεράσουμε τις υποχρεώσεις μας. Το θέμα είναι να ενσωματώσουμε ένα κομμάτι νομοθεσίας μέσα σε μια άλλη νομοθεσία για να αδράξουμε την ευκαιρία που έχουμε για να μειώσουμε τώρα τις εκπομπές αερίων. Για την αξιολόγηση κινδύνου, ναι, η αξιολόγηση κινδύνου όντως ε, χρονολογείται κάποια χρόνια, αλλά η αξιολόγηση αντικτύπου ε, Μιλά για, κάποια, ε, για ένα φάσμα των, ε, του συστήματος ETS. Ε και στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα είμαστε εντός αυτού του φάσματος. Οπότε έχουμε την αξιολόγηση αντικτύπου, μπορούμε να πάρουμε τα, τα αποτελέσματα αυτά, γιατί τελικώς δεν έχει αλλάξει τίποτα για τις τιμές του ETS και το σχετικό φάσμα. Επίσης η Κομισιόν είπε ότι το κόστος για ένα κιλό μπανάνες, ας πούμε, θα αυξηθεί λιγότερο από ένα σέντ. Οπότε δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο τραγικός πια ο αντίκτυπος στους πελάτες ή να μεταφερθούμε από την αυτιλία ας πούμε, στις χερσές μεταφορές επειδή είναι τεράστια η ε, διαφορά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι κίνδυνος αυτό. Και για τα υπόλοιπα που ακούστηκαν, οι εκπομπές στα λιμάνια όντως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα κυρίως σε πόλεις όπου ας πούμε έχει υπάρξει απαγόρευση για τα αυτοκίνητα ντίζελ. Βέβαια μετά δεν άλλαξε τίποτα γιατί ούτως ή άλλως τα πλοία, εκεί που σταμάτησαν να μολύνουν τα αυτοκίνητα, στα... μολύνουν τα πλοία. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία γιατί ακριβώς έχουμε δεσμευτική νομοθεσία για τα λιμάνια που λέει ότι θα πρέπει να δίνουν από, την, από το λιμάνι ηλεκτροδότηση αν υπάρχει ζήτηση. Οπότε τώρα είναι στο, στο χέρι μας να δημιουργήσουμε τη ζήτηση. Αν δεν υπάρχει πλοίο που να ζητά ηλεκτροδότηση από το λιμάνι, γιατί να παρέχει το λιμάνι αυτή τη δυνατότητα, γιατί να επενδύσει σε αυτή την παροχή το λιμάνι. Επίσης, ευχαριστώ τον κύριο Γόλας που ανέφερε το θέμα της, ε, των εκπομπών μεθανίου. Ε, κάναμε, είχαμε μια ενημέρωση χτες, ε, η Επιτροπή Ήτρε, τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε, Δεν είναι ακόμα βεβαίως το πρόγραμμα, αλλά θα το δούμε και ευχαριστώ που το θίξατε, κύριε Γουόλας. Επίσης, κάτι άλλο για αυτά που είπε η κυρία Γιόρντι για τα μέτρα του IMO. Εγώ έχω πάει στον IMO στο Λονδίνο, έχω μιλήσει με άτομα που είτε είναι μέλη του, είτε κάνουν μελέτες για τον IMO. Ο IMO είναι μια υπηρεσία του ΟΗΕ, ένας οργανισμός του ΟΗΕ και έχει κάποιους κανόνες. Οι οποίοι εμένα με εξέπληξαν πρέπει να πω, ας πούμε οι πέντε μεγάλες ε, χώρες ε, σημαίας που είναι υπεύθυνε για πάνω από 50% του φορτίου που μεταφέρεται και έχουν δυνατότητα ε, πλειοψηφίας που μπλοκάρει γιατί και το μεταφερόμενο φορτίο είναι ένα κομμάτι της, της ψηφοφορίας, της διαδικασίας Αυτά τα κράτη σημαία δεν είναι παρόντα ωστόσο στο τραπέζι από μόνα τους ως κυβερνήσεις. Στέλνουν τις ε, ε, εγγεγραμμένες εταιρείε τους. Οπότε η βιομηχανία κάθεται σε αυτό το τραπέζι όταν γίνεται η ψηφοφορία. Οπότε δεν είναι περίεργο που ο IMO δεν έχει προτείνει προοδευτικά μέτρα, γιατί προφανώς τα κράτη-μέλη λένε θέλουμε να γίνεται καταχώρηση στα, κράτη, στα κράτη μας, δεν θέλουμε δεσμευτικά μέτρα για τα πλοία, γιατί αλλιώς θα μπορεί να έχει αυτό αντίκτυπο στις μεταφορές, τις θαλάσσιες και Μπορεί να μην υπάρχουν μεταφορέ από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη και από την Ευρώπη στην Κίνα, α πούμε, που εντάξει, αμφισβητείται βέβαια αυτό. Οπότε ο IMO δεν πρόκειται να προτείνει ποτέ προοδευτικά μέτρα. Είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει αυτή την, ε, αυτό το πρόγραμμα για την ε, μέτρηση της ταχύτητας, γιατί και η ταχύτητα έχει να κάνει με τον ε, θόρυβο και επίσης ο θόρυβος είναι υπεύθυνο για την απώλεια βιοπικιλότητα στη θάλασσα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι θεμητό να το βάλουμε αυτό, είναι συνετό να το βάλουμε αυτό στο MRV. Ίσως καλό θα ήταν να έχουμε δεσμευτικούς ε, στόχους, όπως ας πούμε έχει προταθεί από το Λουξεμβούργο στις αρχές του χρόνου, όταν είπαν ότι έχουμε αυτό το στόχο του 40% και τη μείωση δηλαδή ε, αναμεταφερόμενο ανα φορτίο μέχρι το 2030, γιατί να μην το κάνουμε μόνο Και τελευταίο σημείο, Έχω μιλήσει με κάποιους πλειοκτήτε εδώ τις τελευταίες εβδομάδες, ε, από τη στιγμή που ανάλαβα εισηγήτρια. Πήγα στο Ρότερνταμ την προηγούμενη εβδομάδα σε μια διερευνητική ε, αποστολή, την πράσινη εβδομάδα, και, και μου είπαν ότι έχουμε εφαρμόσει εμεί το σύστημα MRV, γιατί έπρεπε να υποβάλουμε αναφορέ, εκθέσει. Και δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα να, ε, να χρησιμοποιούμε μία παράμετρο, την οποία ούτω ή άλλω γνωρίζουμε. Γιατί προφανώς ξέρουν πόσο, μετα... πόσο φορτίο μεταφέρουν τα πλοία του. Να γράψουν ένα νούμερο παραπάνω μέσα στο, στον... στο Excel δεν είναι τραγικό. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Τουλάχιστον έτσι μου είπαν. Σα ευχαριστώ όλους για την ανταλλαγή απόψεων και βεβαίω προσβλέπω στην σύνταξη της τελικής έκθεσης και Περιμένω και τις τροπολογίες σας. Και περιμένω βέβαια και τη στήριξή σας σε όλα αυτά τα μέτρα που θέλουμε όλοι να δούμε να εφαρμόζονται μέσω αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Thank you. Can applaud if you like. <laughs> okay. So it was the... Αυτή ήταν η πρώτη πρώτη συζήτηση για αυτό το θέμα. Έχουμε ε, τη συζήτηση του σχεδίου έκθεση το Φλεβάρι. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών το Μάρτιο. Εδώ θα ψηφιστεί το Μάιο η έκθεση αυτή. Έτσι έχουμε προγραμματίσει. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Λαθρεμπόριο ζώων συντροφιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφορική ερώτηση. Θα δώσω το λόγο ε, τον κύριο Σπόσλακ, εκπρόσωπο του ΕΛΚ, για να ε, κάνει την πρώτη παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα βάλω τα δυνατά μου για να είμαι σύντομος, γιατί ξέρω ότι στις 12 έχουμε ε, αυτή την πανηγυρική εκδήλωση που πρέπει να πάμε, την υπογραφή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει πάρα πολλά ε, για τα ζώα στην Ευρώπη αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά που μπορούν να βελτιωθούν πάντα υπάρχει το καλύτερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα εκτεταμένο λαθρεμπόριο ζώων συντροφιάς. Αυτό το λαθρεμπόριο είναι πολλές φορές και εξαιρετικά επικερδές. Υπάρχουν διαφορές βέβαια μεταξύ κρατών μελών ως προς την ευημερία και αυτό καθορίζει και τις τιμές και υπάρχουν διαφορές στις τιμές. Και ε, αυτό το εκμεταλλεύονται διάφοροι απατεώνες ε, για να ε, κάνουν αυτό το λαθρεμπόριο ζώων συντροφιάς, τα οποία μεταφέρουν από χώρα σε χώρα και καμιά φορά οι σκύλοι και οι γάτες ζουν πραγματικά δράματα. Ε, τα έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια ε, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και χάρη σε κάποιους δημοσιογράφους της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ρεπόρτερ, ξέρω ότι η κατάσταση είναι διαδεδομένη σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ε, με τις συνθήκες διαβίωσης ε, των ζώων και την ευημερία τους, αλλά είναι και οικονομικό. Έχει να κάνει με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, τη εσωτερική αγορά, την προστασία των καταναλωτών, την απώλεια φορολογικών εσόδων και άλλες ε, ολέθριες συνέπειε αυτή της παράνομη δραστηριότητα. Δυστυχώς, ε, πολύ συχνά ο κόσμος βρίσκεται σε πλήρη άγνοια για το τι τραβάνε τα ζώα συντροφιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό υπάρχει ανάγκη να κάνουμε ε, ένα πρώτο βήμα. Ε, να καταγράφουμε, να κάνουμε μια απογραφή των σκύλων και των γάτων. Ε, και στόχος της πρότασης λοιπόν είναι να ζητήσει επιγόντως από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμιστεί αυτό με τις κατεξουσιοδότηση πράξης και λοιπά, να έρθει μια πρόταση για μια μέθοδο με την οποία να καταγράφονται και να ταυτοποιούνται οι σκύλοι και οι γάτες σε βάσεις δεδομένων των κρατών μελών. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι βάσεις δεδομένων να είναι ε, συμβατές μεταξύ τους και να υπάρχει διαλειτουργικότητα ε, και ε, με τα διαβατήρια των ζώων συντροφιάς. Έχω και κάποιες τροπολογίες να προτείνω και πραγματικά ελπίζω να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να βελτιώσουμε τη ζωή των ζώων συντροφιά Από τους Σοσιαλιστέ και δημοκράτε, η κυρία Σπούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η προστασία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωση και των δικαιωμάτων των καταναλωτών ενάντια στις αρνητικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου ε, από το εμπο... Ε, ζώων, καθώς και η προστασία της ε, ευημερία των ζώων είναι πολύ σημαντικές. Καλούμε την Κομισιόν, λοιπόν, να προτείνει αυστηρότερου κανόνε για την καταγραφή των σκυλιών και γατιών για να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο. Θα πρέπει αυτές οι βάσεις δεδομένων να είναι συνδεδεμένες στα κράτη-μέλη. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε το εμπόριο αυτό γιατί είναι γύρω στο 80% του συνόλου του νόμιμου εμπορίου. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν λοιπόν να φτιάξει ένα διατομεακό πρόγραμμα δράσης για την Ένωση ώστε να επιβληθούν αυστηρότερες ποινές, καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία στην επιβολή του νόμου, επιπλέον αυστηρότεροι κανόνες και απαιτήσει για την υγεία και ευημερία των ζώων. Χρειάζεται χρειάζεται κατάρτιση για την επιβολή του νόμου, καθώς και εκστρατείε για να ε, ε, αυξηθεί η ενημέρωση για τους δυνητικού ε, αγοραστές. Θα υποβάλω τροπολογίε για να καταστήσουμε το ψήφισμα πιο ισχυρό χρειάζεται να επιβληθεί αυστηρότερη ε, ε, προθεσμία για την Κομισιόν ώστε να υιοθετήσει γενικά τα μέτρα. Ε, από την άποψή μας θα πρέπει οι online πολιτές να περιορίζονται από, από απαιτήσει ώστε να περιοριστεί το επιγραμμικό εμπόριο ζώων. Έτσι θα προστατεύσουμε τα ζώα και την ευημερία τους. Ευχαριστώ πολύ. Από το ο κύριος Χότσικ. Είναι ένα από τα θέματα που με έχει απασχολήσει πολύ καιρό γιατί εργάστηκα σε οργανισμούς προστασίας ζώων, ιδιαίτερα ε, αυτό που το οποίο υποφέρουν ε, τα ζώα, είναι, μάλλον τα ζώα τα οποία υποφέρουν περισσότερο είναι τα σκυλάκια, τα κουταβάκια. Ε, ιδιαίτερα στη Σλοβακία ε, δεν υπάρχει ε, πολύ έλεγχος. Δεν είναι μόνο τα ζώα που υποφέρουν, είναι αθώα ζώα, αλλά αφορά το θέμα και την ανθρώπινη υγεία, ε, γιατί μπορεί τα ζώα αυτά να μεταφέρουν ε, κάποιες αρρώστιες όταν είναι παράνομο το εμπόριο, αλλά έχει και να κάνει με το κράτος δικαίου, ότι το παράνομο εμπόριο ζώων είναι μεγάλο κομμάτι του λαθρεμπορίου και επίσης έχει να κάνει και με την ψηφιακή αγορά γιατί οι επιγραμμικέ πλατφόρμες τη σήμερα ημέρα παίζουν μεγάλο ρόλο στην εμπορία ε, ζώων συντροφιά. Δεν υπάρχουν πια τα pet shop, τα καταστήματα ε, όπου μπορεί κανείς να αγοράσει ζωάκια αλλά τα περισσότερα κυκλοφορούν μέσω του ίντερνετ. Αν έχουμε σωστή εφαρμογή του νομοθεσία περί υγείας των ζώων με διασύνδεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και όλα αυτά συνδέονται με την, τις επιγραμμικές πλατφόρμες, μπορούμε πραγματικά να περιορίσουμε το παράνομο εμπόριο πολύ χωρίς μεγάλο φόρτο για κανέναν, γιατί υπάρχουν εθνικά συστήματα καταγραφής ε, σε όλα τα κρατη Ελπίζω λοιπόν πως ε, θα περάσουν αυτά όλα και θα δούμε όχι μόνο απαντήσεις προφορικές αλλά και συγκεκριμένε δράσεις από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλιπς, ε, εξ ονόματος των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη ανθίζει η ε, εκτροφή σκύλων και γατιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 60 εκατομμύρια σκύλοι και 64 εκατομμύρια γάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπολογιστεί ότι κυκλοφορούν. Τώρα πόσο ακριβείς είναι αυτές οι υπολογισμοί δεν το ξέρουμε γιατί δεν λειτουργεί σωστά και δεν γίνονται πλήρως ε, η αναγνώριση και ο εντοπισμός ε, και η καταγραφή των ζώων. Δεν υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στις εθνικές και περιφερειακές βάσεις και δεν υπάρχει καμία υποχρεωτική ε, ρύθμιση για την καταγραφή των ζωών συντροφιάς. Αυτό ανοίγει το δρόμο για παράνομους εμπόρους αλλά και εκτροφή παράνομη ε, και αυτό επιφέρει βλάβη στην ευημερία και υγεία των ζώων που πολλούνται αλλά είναι και απειλή για τη δημόσια υγεία, την προστασία των καταναλωτών, τη διαχείριση των πληθυσμών αδέσποτων και την συμπεριφορά υπεύθυνων ε, ιδιοκτητών ζώων συντροφιά. Εγώ είμαι ευτυχής που βλέπω αυτό το ψήφισμα, ιδιαίτερα γιατί καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για σύμμορφα και ε, αλληλοσυνδεόμενα συστήματα σε όλα τα κατημέλη. Όμω, θα ήθελα να προχωρήσουμε και περισσότερο και να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε υποχρεωτική αναγνώριση, ταυτοποίηση σκυλιών και γατιών που θα πρέπει να γίνεται από του πολιτέ πριν αγοραστούν ε, για πρώτη φορά τα ζώα αυτά, καθώς και πιο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τον κανονισμό για το εμπο... τη ρύθμιση μάλλον του εμπορίου ε, από επιγραμμικές πλατφόρμες. Θα συνεργαστώ με τους εκπροσώπους των άλλων ομάδων για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. ID. Η κυρία ε, Μπρούνα. Ε, συνέπειες δραματικές υπάρχουν για τα ζώα, τα οποία εκτρέφονται και μεταφέρονται σε απαραίτητες συνθήκες ε, και υπόκεινται πολύ ε, κακή διαχείριση, αλλά είναι και πολύ, θέμα, πολύ μεγάλο θέμα υγείας όσον αφορά τη διάδοση ασθενειών όπως η λύσα. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχονται τα ζώα και οι άνθρωποι, ακόμα και όταν είναι νόμιμο το διασυνοριακό εμπόριο ζώων, είναι θύμα dumping, όπου διαρκώς μειώνονται τιμές και αυτό γίνεται εις βάρος των ζώων. Το μεγαλύτερο αίτιο για το παράνομο εμπόριο και την ε, ε, και, την πλαστοποίηση των στοιχείων των ζώων είναι ακριβώς ε, αυτό που οδηγεί ε, ειδικά στο εμπόριο στην, ε, στις, σε κάποιες από τις ανατολικές χώρες της Ένωσης γιατί γίνεται και εκτροφή από μία επαγγελματίε. Επίσης θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτά τα εργοστάσια κουταβιών τα οποία λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο η πώληση δε των ζώων επιγραμμικά θα πρέπει να αφορά μόνο τους επαγγελματίες εκτροφής και τους ε, ε, ε, ιδιώτες που αναπαράγουν τα ζώα τους μόνο και μόνο λόγω της αγάπης που φτρέφουν γι' αυτά και θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρά ρυθμισμένο πλαίσιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ καλωσορίζουν αυτό το ψήφισμα για το παράνομο εμπόριο ζών συντροφιά. Θα ήθελα να πω <coughs> ότι η ECR έχει υποβάλει αυτό το ψήφισμα ήδη τον Ιανουάριο του 2018, αλλά δυστυχώς δεν μπήκε σε ψηφοφορία. Χαίρομαι που μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτή τη θητεία τη δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα και ελπίζω να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί από το προηγούμενο κοινοβούλιο. Ε, το εμπόριο ε, ζώων και η έλλειψη ε, νομοθετικού πλαισίου προφανώς δημιουργεί επιπλοκές και αρκετά προβλήματα για την ευημερία των ζώων. Η πώληση ζώνων συντροφιάς από το ίντερνετ είναι ένα κομμάτι της λειτουργίας της ε, ε, ενιαίας αγοράς. Υπάρχει ε, απώλεια εσόδων, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Πολλοί κανόνες καταπατούνται. Αυτό λοιπόν το σχέδιο ψηφίσματος λαμβάνει πολλές από τις δικές μας παρεμβάσεις του εγγράφου του 2018 και θα πρέπει να ζητήσουμε την υιοθέτηση κατοξιώδηση πράξεων που θα προβλέπουν ένα λεπτομερές και συμβατό σύστημα για την ταυτοποίηση των ε, γατιών και των σκυλιών, χρησιμοποιώντας πάντα τις βάσεις δεδομένων που έχουν τα κρατη Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν και διατομεακά σχέδια δράσης μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να ε, υπάρξουν επίσης πιο σοβαρά και πιο αυστηρά πρόστιμα και πρέπει να υπάρξει και καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Θα υποβάλω εγώ κάποιες ε, τροπολογίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μένα και θα ήθελα το έγγραφο αυτό να είναι υψή τη Και βεβαίως Προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους συνσηγητές. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, τα είπαν όλοι. Μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα, το λαθρεμπόριο σε ζώα, ε, ιδιαίτερα σε σκυλιά και η γατιά, είναι από τις πιο κερδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη για τα κουτάβια που είπατε εσείς, κυρία μου. Από την Ανατολική Ευρώπη ε, ε, έρχονται στη Δυτική Ευρώπη και αυτό σημαίνει τρομερά βάσανα. Πολλά ε, αρρωσταίνουν, πολλά απογαλακτίζονται πάρα πολύ νωρίς και μετά έχουν προβλήματα στη συμπεριφορά. Ας πούμε στην Ολλανδία πολιούνται με τρόπο απατηλό ε, ηλεκτρονικά. Δεν γίνονται σωστοί οι εμβολιασμοί ε, και αυτό είναι κίνδυνος και για τον ιδιοκτήτη. Δεν είναι μόνο η λύσα, υπάρχουν και άλλες αρρώστιες που μεταδίδονται, όπως είναι η λαϊσμανίαση. Υπάρχει υποχρέωση στην Ευρώπη να, να, να έχουν διαβατήρια και ηλεκτρονικό τσιπ. Αλλά πολλέ φορές παστογραφούνται όλα αυτά τα στοιχεία και στο τσιπάκι δεν μπαίνει αρκετή πληροφορία. Στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστε απαιτήσει γιατί τι θα έχει αυτό το ηλεκτρονικό τσιπάκι. Α πούμε, ε, τα στοιχεία του εκτροφέα, του μεσάζοντα, του ιδιοκτήτη. Να υπάρχει ε, η δυνατότητα αντιμετώπιση όχι μόνο του λαθρεμπορίου, αλλά της κακομεταχείρισης των ζώων. Κοιτάξτε τι φρικτά συμβαίνουν ε, με τα ε, σκυλιά γκάλγκο στην Ισπανία. Καλά, δεν θα σου πω τώρα τις αφρικαστικές αυτές λεπτομέρειες, αλλά πολλές φορές ε, πολλοί διοκτήτες τέτοιων σκυλιών πιστεύουν ότι όσο περισσότερο κάκο μεταχειρίζονται και βασανίζουν το ζώο, τόσο καλύτερες επιδόσεις θα έχει στο κυνήγι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να, μην τα αφήσουμε στην άκρη. Αυτό να το συμπεριλάβουμε. Στο ψήφισμα επίσης γίνεται λόγος για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των κουταβιών με καλύτερο τρόπο ανείχνευσης και αντιμετώπισης. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με αυτές τις φρικαλαιότητες, ε, να το κάνουμε κτήμα μας για να τερματίσουμε και τα βάσανα αυτά των ζώων, αλλά και τη διάδοση ασθενειών από τα ζώα συντροφιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν έχουμε χρόνο τώρα για κάτι και τέτοια, οπότε θα δώσω αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρία λεπτά από τη Γενική Διεύθυνση ε, Υγείας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Όντως ε, δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη. Πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας ενημερώσω για το τι κάνει η DG η Σαντέ Υγείας για αυτό το σημαντικό τομέα. Και θα ξεκινήσω αναφέροντας τις νομοθετικές πτυχές. Ε, κάναμε refit στις νυφιστάμενες ε, οδηγίες 9265 που ασχολείται με το εμπορικά ζητήματα για τα ζώα συντροφιάς αντικαθίσταται και ε, αναθεωρείται από την ε, νομοθεσία περιγείας των ζώων από το 2021, πρώτη πρώτου 2021. Ε, Επίση, ε, η 576 του 2014 θα περιληφθεί στον ίδιο νομοθεσία, αλλά θα ισχύσει ε, μεταβατικά μέχρι το 2026. Άρα, λοιπόν, το αίτημα για αναθεώρηση έχει γίνει για την οδηγία 9265 και για την 576 του 2014 που σχετίζεται με τη μη εμπορική κίνηση ζώων, μετακίνηση ζώων, γιατί αυτή ήταν η απόφαση των συνομοθετών όταν συνέταξαν την νομοθεσία περιγείας των ζώων. Για να τονίσω τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας νομοθεσίας για την υγεία των ζώων, καθώς και των κατεξοδότηση πράξεων που θα ισχύσουν από τον Απρίλιο του 2020, 2021 θέλω να τονίσω κάποια στοιχεία που σίγουρα θα σας βοηθήσουν. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως η νομοθεσία περιγείας των ζώων ορίζει υποχρεωτική καταγραφή των ε, καταστημάτων που, για εκτροφής ε, ε, σκύλων και γάτων. κατά, κατά εξοδότηση δε πράξη εισάγει δύο νέα στοιχεία όπως η υποχρεωτική καταγραφή των μεταφορέων που μεταφέρουν σκύλους και γάτες ανάμεσα στα κρατη και επίσης σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες. Επίσης έχουμε ε, υποχρέωση έγκρισης για τα καταφύγια και ε, από τα οποία θα μετακινηθούν αυτά τα ζώα ανάμεσα στα κράτη-μέλη και βεβαίως υπάρχει και υποχρέωση για ε, καταγραφή των ε, ζώων συντροφίας όταν μετακινούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις λοιπόν για να βελτιωθεί ε, η, καταγραφή, η ταυτοποίηση και η ανιχνευσιμότητα των ζώων συντροφιάς και αυτό περιλαμβάνει και την καταγραφή των κουταβιών όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο του ψηφίσματός σας και των εκτροφέων για να βελτιωθεί η, ο έλεγχος. Επίσης, Επίσης συντάσσεται νέα της πράξη με πρόταση για λεπτομερή και συμβατά συστήματα για του τρόπου και μέσα ε, εντοπισμού ε, καταγραφής ε, το, σε βάση δεδομένων των κρατών μελών που θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένες. Πριν λοιπόν αναλυφθεί τέτοιο μέτρο θα πρέπει να γίνει ένα, μια μελέτη αντικτύπου και αυτό για να φανεί και αν υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ελέγχου παράνομου εμπορίου ε, σκυλιών και ε, γατιών. Εμείς εστιάζουμε λοιπόν στην ανάπτυξη των συστημάτων που χρειάζονται για να υλοποιηθεί σωστά αυτό το σύστημα. Τώρα όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας που επίσης αναφέρθηκε με χαρά να σας πω ότι ενεργούμε σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διάφορες ε, σε διάφορους τομείς. Πρώτον, ε, ε, ελεγκτικός κανονισμός ε, μας οδήγησε στην έναρξη του προγράμματος συντονισμένου ελέγχου του 2018 για τον έλεγχο των αδέσποτων σκυλιών και γατιών με τους εξής στόχους. Να βοηθήσουμε... Μπορείτε να ολοκληρώσετε παρακαλώ. Διακόπτει ο Πρόεδρος, μπορείτε να κλείσετε την παρέμβασή σας παρακαλώ. Μάλιστα. αναφερόμουν στην επιβολή Κοιτάξτε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, μπορείτε να ολοκληρώνετε την παρέμβασή σας. Μάλιστα, Πρόεδρε. Το, το ολοκληρώνω λέγοντας πως έχουμε ήδη προτείνει μέτρα στον τομέα της, υγείας, το, της νομοθεσίας περί υγείας των ζώων. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κρατημέλη ώστε να βελτιώσουμε την ε, επιβολή όχι μόνο των σχετικών νομοθεσιών αλλά και στο πλαίσιο της πλατφόρμας για την υγεία των ζώων και επίσης όσον αφορά την κατάρτιση και συνεργασία των κρατών μελών, ήδη από το 2013 εργαζόμαστε στο πλαίσιο του, της ασφαλέστερης ε, ζωοτροφής με τους, μαζί με το κτηνιατρικό συμβούλιο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας. Οι ψηφοφορίες θα γίνουν ε, το απόγευμα και για το ψήφισμα υποβολή ε, τροπολογιών θα, γίνει στις... θα είναι στις 12 Νοεμβρίου στις, 12 το μεσημέρι. Και αυτά. Ε, στόχος να περάσει από την Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Περνάμε στο τελευταίο σημείο που έχουμε πριν από την ε, τελετή έμας ε, προφορική ερώτηση και ψήφισμα για τη διευκόλυνση, για τη ψηφιακή μετάβαση, για την υγεία και την ασφάλεια, ώστε να φτιάξουμε μια ε, κοινωνία όπου η υγεία θα έχει την προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο στον κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλούμε για την ψηφιακή ενιαία αγορά που προωθεί την υγεία του πληθυσμού, την ίση πρόσβαση στην περίθαλψη και την σωστή χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων. Το ερώτημα είναι πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαχειριστεί αυτή την ψηφιακή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, του τομέα της υγείας. Γιατί το θέμα δεν είναι απλώς να κάνουμε καινοτομίε για να τις κάνουμε. Μιλούμε για συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των περιφερειών, συνεργασία με, τη, με τα σχολεία, έτσι ώστε να καταδεικνύεται και η προστιθέμενη αξία του εγχειρήματο και βεβαίω μιλούμε για τη βελτίωση τη εργασία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να πω συγγνώμη στην κυρία Εύη. Ξέχασα να σας δώσω το λόγο στην προηγούμενη συζήτηση ως μία εγγεγραμμένη. Δεν σας είχα στον κατάλογό μου. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στο θέμα. Σέρδας. Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές προκλήσεις Έχουμε και την επιδημιολογική μετάβαση, όπου οι πολίτε ε, ζουν μεγαλύτερα για περισσότερα χρόνια και επίση έχουμε τι μη μεταδεδόμενε ασθένειε. Ε, αυτές οι προκλήσει είναι σημαντικέ για τα συστήματα υγεία και υπάρχει ανάγκη για ψηφιακέ λύσει που θα προωθούν την υγεία, θα προβλέπουν τι ασθένειε και θα επικεντρώνονται στον ασθενή και στι ανάγκε του για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν έχουν τη δυνατότητα να, να, γίνει, να κάνουμε αυτή την ψηφιακή, το ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς, τη βοήθεια των κρατών μελών και οι πολίτες ακόμα δεν μπορούν να υποφεληθούν ε, πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν λοιπόν αυτές οι εξελίξεις ε, για την, για πολιτικές υγείας με βάση αποδεκτικά στοιχεία για τις μεταδεδομένες ασθένειες και για την έγκαιρη πρόγνωση των ε, απειλών για τη δημόσια υγεία. Η πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να ε, είναι εγγυημένη και η κυβερνοασφάλεια επίσης για να μειώσουμε τον κίνδυνο των ε, παραβιάσεων της ιδιωτικότητας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχουμε την εφαρμογή του κανονισμού GDPR. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τα συστήματα και τη διαλειτουργικότητά του μεταξύ των διαφορών μητρών και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι απαραίτητη, καθώ επίση και η κατάρτιση του εργαζομέ... των εργαζομένων στον τομέα τη υγεία πρέπει να έχουν τι απαραίτητε δεξιότητε και τα προσόντα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τέλο, η ψηφιακή υγεία έχει τη δυνατότητα να ε, βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες υγείας, την παροχή αυτών στους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να έχουν ε, βεβαίως ε, και την γνώση για να μπορούν να έχουν υγιείς συνήθειες και να προωθούν τις στρατηγικές υγείας πρέπει βεβαίω να εξασφαλίσουμε και την προσβασιμότητα. Ζητούμε αυτέ οι προτάσει να συμπεριληφθούν στην πρόταση για, την, για το ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για την Υγεία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για δεύτερη φορά συζητούμε αυτό το ψήφισμα. Ήδη είχαμε εργαστεί πριν από ένα χρόνο σχεδόν ακριβώς ε, με αυτό το θέμα. Οι εκλογές μας ε, εμπόδισαν από το να το ψηφίσουμε στην Ολομέλη. Παραμένει το μήνυμα το ίδιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ε, για να συνοδεύσουμε την ψηφιακή μετάβαση ε, των υπηρεσιών υγείας. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το νοσηλευτικό προσωπικό. Ε, ας πούμε κάθε πότε πρέπει να παίρνει το φάρμακό του ένας ασθενής, να μετράει το ζάχαρο του ή ακόμα και να εντοπίζουμε γεωγραφικά ασθενείς που έχουν κάποια διανοητική σύγχυση. Ε, σε αυτά ε, θα ήθελα να επιμείνω στις αρχές μας και στο μήνυμά μας. Η προτάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο ψήφισμα θελήσαμε να επιμείνουμε σε τρία βασικά για μας σημεία. Ε, οποιοδήποτε επιγραμμικό σύστημα θα πρέπει να είναι θωρακισμένο από πλευράς ασφάλειας ηλεκτρονικής. Είμαστε εδώ αδιάλακτοι. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε για τα ευρωπαϊκά συστήματα, δηλαδή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να εγγυηθούμε τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, των δεδομένων με εναρμόνιση ε, των ε, τύπων που μας ζητούν όλοι οι χρήστες και το τελευταίο που είναι και ακρογωνιαίος λήθος θα πρέπει ε, να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται στη συνέχεια όλοι οι χρήστες, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, γιατροί, όλες οι ειδικότητες. Επίσης θα κάνω μια τροπολογία για να προσθέσω το εξή. Θα πρέπει να προβληματιστούμε ε, ως προς τη διοντολογική διάσταση αυτής της ηλεκτρονικής επανάστασης στις υγειονομικές υπηρεσίες. Μέχρι πού επιτρέπεται οι αλγόριθμοι να παίρνουν αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη επέμβαση. Είναι πάντα ουδέτερα τα δεδομένα. Μόλις ανακαλύφθηκε στις Ηνωμένε ότι έχουν βάλει κριτήρια, όχι ο αλγόριθμος, από τα δεδομένα που δίνουν ε, φιλετικά για να δουν ποιους θα ε, ε, θεραπεύουν κατά προτεραιότητα. Ο πληθυσμός γερνάει, είναι όλο και πιο απαιτητικοί ασθενείς και καλά κάνουν. Έχουμε τις δυνατότητες τώρα τις ψηφιακές να τους διευκολύνουμε την πρόσβαση και να βελτιώσουμε πολύ την ποιότητα ζωής τους και στο τέλος της ζωής τους. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα ναι στην ηλεκτρονική αυτή επανάσταση, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Αυτό ζητούμε από την Κομισιόν στο ψήφισμά μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Όκεν από τους Πρασίνους. Øh, Θα μιλήσω δανέζικα, Πρόεδρε. Κάναμε μια πολύ έντονη συζήτηση στην Δανία για τα θέματα αυτά. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στο ε, προβληματική του θέματος, γιατί έχουμε έναν ε, πολύ μηχανικό φιλελευθερισμό για το τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί κίνδυνοι τους οποίους θέλω να αναφέρω. Ε, ένας από τους στόχους είναι να φύγουν οι γιατροί από την προσφορά ε, υπηρεσιών στους ασθενείς. Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Η επαφή μεταξύ του ιατρού και του ασθενούς είναι ζωτική σημασίας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό μόνο και μόνο για να εξοικονομήσουμε πόρους. Επίσης, υπάρχει υψηλό επίπεδο ε, ψηφιακής αγραμματοσύνης. Ε, όχι μόνο στις, στις χώρες του τρίτου κόσμου και στις πλούσιες χώρες. Πολλοί κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και δεν είναι θέμα αν είναι νέος ή αν είναι ηλικιωμένος. Είναι θέμα κοινωνικών τάξεων και πώς αυτές έχουν διαφορετική πρόσβαση σε αυτές τις ψηφιακές λύσεις. Οπότε χρειάζεται καλύτερη εξοικείωση όλων με τον τομέα αυτό, έτσι ώστε και οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός GDPR θα εφαρμοστεί πλήρως πόρο απέχουμε από το να συμβεί αυτό. και μπορεί απλώ να είναι αέρας φρέσκο αυτά που λέμε, ότι σεβόμαστε τον GDPR κτλ. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι ω προ αυτό. Και για να κλείσω, να πω ότι θα ήθελα να προειδοποιήσω για κάτι. Τα δεδομένα για την υγεία είναι τα πιο ε, πολύτιμα δεδομένα και μοιράζονται παντού. Και λέμε εδώ πολύ χαλαρά ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν όλα τα ιατρικά δεδομένα, να αποθηκεύονται εδώ και εκεί. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο για το καλό της υγείας μας, γιατί αλλιώς θα έχουμε σημαντικά προβλήματα. Τίποτα δεν είναι δωρεάν άλλωστε. Και όσοι από εμά δουλεύουμε με τέτοιες ψηφιακές ε, λύσεις και βλέπουμε πόσα ε, κονδύλια παίζονται, ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Το θέμα δεν είναι απλώς να έχουμε συστήματα υγείας και πιο αποτελεσματικά και πιο ασφαλή. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την τεχνική, πρέπει να είμαστε πολύ πιο ε, υποψιασμένοι για αυτή την ε, τεχνολογία. Ευχαριστώ. Για την ECR, η Ιωάννα Κοψίνσκα. Κοψίνσκα, mm, Πρόεδρε. Mm. Ε, ευχαριστώ. Η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των μελλοντικών συστημάτων υγείας του, είτε σε επίπεδο εθνικό, κρατών μελών, είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το Τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι, είναι αυτή η σωστή χρονική στιγμή για να μιλήσει κανείς για πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα. είναι ώρα επιτέλους να αρχίσει μια συζήτηση για αυτό και εγώ υποστηρίζω πλήρως οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να επιτρέψει ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα. Αλλά θα ήθελα να δω και επίσης ε, υψηλής ποιότητος δεδομένα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερη φροντίδα με κέντρο των ασθενή, να βελτιώσουμε την υγεία των πολιτών και όντως να βασίσουμε την προσέγγιση μας στον ασθενή. Πολλά μπορούν να γίνουν ακόμη και σε επίπεδο κράτους μέλους αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω το κείμενο του ψηφίσματος και υποστηρίζω τα όσα υπόθηκαν για την προσέγγιση με βάση τον ασθενή και βεβαίως την προσέγγιση την ολιστική, τη συνολική που είναι σωστή κυρίως υπό το φως όλες τις συζήτησεις που γίνεται για την πρόσβαση στα δεδομένα ε, και μπορεί να υπάρξουν ε, θερμές συζητήσεις ε, υπάρχουν φωνές που λένε, που μιλούν για την κυβερνοασφάλεια κτλ. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο ο ασθενής το θέμα είναι το σύνολο των δεδομένων που υπάρχουν στο ίντερνετ. Μία νέα πολιτική ολοκληρωμένη για την υγεία είναι ιδιαίτερος σημαντική και τα δημόσια συστήματα υγείας είναι, έχουν να παίξουν ρόλο και στην ε, μετάβαση στην ψηφιακή υγεία. Επίσης καλωσορίζουμε την αναφορά στην δήλωση και την ιδέα ενός νέου παραδείγματος για την υγεία που βεβαίως σχετίζεται πάντα και με το ε, υψηλό κόστος. Η παράγραφος 16 μιλάει για τις συστάσεις του, ε, της ΠΟΗ. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι το σημείο κλειδί και θα χρειαστεί βεβαίως σημαντική συζήτηση. Ε, διακόπτει ο πρόεδρος, μπορείτε να ολοκληρώσετε. Ένα λεπτό, λέει η κυρία Κομπτσίνσκα. Ε, ολοκληρώστε παρακαλώ. Η μετατροπή που βλέπουμε να γίνεται χρειάζεται ε, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή τη νέα καινοτόμα τεχνολογία και να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Η Πολωνία εμπλέκεται στην καινοτομία, στην κατάρτιση, εκπαίδευση. Και έχουμε δει ε, γιατρούς ε, που είναι και μέχρι και 70 χρονών και παρόλα αυτά ε, χρησιμοποιούν, ε, στέλνουν ηλεκτρονικές συνταγές. Για την ΚΟΕ η κυρία Κονέτσνα δεν είναι εδώ. Ωραία, να ακούσουμε την Κομισιόν για ένα λεπτό περίπου και μετά θα έρθει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η Κομισιόν ε, είναι προσιλωμένη στην πρόθεση της ψηφιακή ε, μετάβασης όπως έχει αυτό αναφερθεί στην ανακοίνωση του 2018 για την ε, συμπερίληψη της υγείας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ανακοίνωση αυτή είναι δομημένη σε τρεις πυλώνες. Καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στην ε, ασφάλιση των δεδομένων. Καλύτερη, το δεύτερο είναι η καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα για να προωθηθεί η έρευνα και η προσωπική, η ατομική, ε, η υγειονομική περίθαλψη. Και η τρίτος είναι ε, οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας. Σε αυτό το τομέα συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και έχουμε ήδη πετύχει πρόοδο σε, στους τρεις αυτούς τομείς, αλλά η Κομισιόν επίσης γνωρίζει τι ε, κρεμεί ζητήματα και τις προκλήσεις ε, και θέλει να δουλέψει περισσότερο για τα θέματα που περιγράφονται στο α, ανακοίνωση του 2018 σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και αυτό τονίστηκε και από τον υποψήφιο Επίτροπο για την Υγεία. Δημιουργία δηλαδή ενός χώρου, ευρωπαϊκού χώρου ε, δεδομένων υγείας. Μάλιστα. Και εδώ ολοκλήρωσα την παρέμβασή μου. Okay, thank you. We are on time. Ακριβώς την ώρα μας. I'm going to switch to French. Θα τα πω γαλλικά. Pour accueillir euh, Euh, για να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, την Αντιπρόεδρο και τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Στη μεγαλύτερη σήμερα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σημαντικότερη. Ε, φαίνεται το ενδιαφέρον των μελών και της ε, κοινοβουλευτικής ε, αυτής θητείας για τα θέματα περιβάλλοντος. Ήρθατε εδώ στην Επιτροπή για να υπογράψετε τις δεσμεύσεις και τις, ε, τα όσα έχει υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί καλό είναι να δίνουμε μαθήματα για το περιβάλλον στους άλλους και ακόμα καλύτερο να ε, κάνουμε εμείς τα καθήκοντά μας. Πριν την επίσημη υπογραφή του συστήματος ΕΜΑΣ, του Περιβαλλοντικού του Κοινοβουλίου, θα μας πείτε τι καταφέραμε συλλογικά, βέβαια τα μέλη και οι υπηρεσίες, το προσωπικό, αλλά και προς τα που θα πρέπει να κινηθούμε. Γιατί αν θέλει να αυξήσει τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και το υποστηρίζουμε περισσότερη κυκλική οικονομία, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, θα πρέπει εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας ως Κοινοβούλιο, να ενισχύσουμε τους δικούς μας στόχους για να είμαστε εις το ύψος των διακυβευμάτων. Σας δίναμε στο λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ Προέδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ναι, πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Αυτό είναι ε, το νόημα όλων αυτών. Γιατί Έχουμε ένα, ένα κοινοβούλιο που νομοθετεί για τους άλλους, ζητεί την καλή συμπεριφορά των υπολείπων και φυσικό είναι να πρέπει να δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο Χάουταλα και όλους εσάς για την δέσμευσή σας. Γνωρίζετε ότι από το Δεκέμβριο του 2007 το Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει αυτό το σύστημα διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου στις τρεις έδρες εργασίας εργασίας του σύμφωνα με τον κανονισμό εμάς. Η σημερινή καταγραφή του Κοινοβουλίου ισχύει μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 και είναι υπό εξέλιξη εργασίες για την ανανέωση αυτής της εγγραφής και τα αποτελέσματα του τελευταίου ελέγχου του, του Κοινοβουλίου για το σύστημα ΕΜΑΣ είναι πολύ θετικά και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών θεσμών που εγγράφηκε στο ΕΜΑΣ το 2007 και έχει σήμερα ένα από τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που είναι τα πιο όρημα και τα πιο προηγμένα από όλους, όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό χάρη στην λειτουργία αυτής ε, της ε, εφαρμογής του εμάς εδώ και πάνω από δεκαετία. Είχαμε λοιπόν μείωση 37,7% των εκπομπών άνθρακα, διεξιδίου του άνθρακα του το 2018 σε σύγκριση με το 2006. Σημαντική μείωση κατανάλωσης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση 60% στην κατανάλωση χαρτιού σε σύγκριση με το 2006. 23% μείωση των, ε, των ε, της πατάλης τροφίμων και αύξηση του ποσοστού ε, ανακύκλωσης των αποβλήτων ε, της τάξης 70%. Σημαντικά αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει σε αυτά να, να σταματήσουμε. Με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα γίνεται μια ανταλλαγή εμπειριών ε, με κάποια εθνικά κοινοβούλια που τώρα φτιάχνουν συστήματα διαχείρισης, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ξεκινούν την πορεία τους προς την εγγραφή του στο σύστημα ΕΜΑΣ. Είμαστε λοιπόν σημείο αναφοράς για πολλούς θεσμούς, όχι μόνο ευρωπαϊκούς αλλά και εθνικούς. Της 17 Σεπτεμβρίου, 16 Σεπτεμβρίου 2019, το ξέρετε, το Προεδρείο υιοθέτησε τη νέα περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση του θεσμού μας να διατηρήσουμε την εγγραφή μας στο ΕΜΑΣ βεβαίως, αλλά και να συνεχίσουμε την περιβαλλοντική μας προσέγγιση και διαρκώς να τη βελτιώνουμε. Είμαι ότι η νέα πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική αυτή θα δώσει μεγαλύτερη όθηση στο Ευρωκοινοβούλιο και στις καινοτομίε, στις δημιουργικές ιδέες, στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, ενώ θα εξασφαλίζουμε την εφαρμογή στην πράξη αυτά τα οποία εμείς διακηρύσουμε στους άλλους, δίνοντας έτσι το καλό παραδείγμα. Δεν έχουμε λοιπόν δεύτερο πλανήτη και άρα ο καθένας από εμά θα πρέπει να παίξει το ρόλο του. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τη δική σας προσήλωση, για την προσπάθεια που κάνατε και εσείς ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Dobbiamo firmare.